ασκεί επικοδομητική δουλειά προτείνοντας λύσεις. Δουλειά που ελπίζω ότι εμείς θα ολοκληρώσουμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τις ε, θέσεις της Κομισιόν και να βελτιώσουμε και την ποιότητα της πρότασης. Εγώ ελπίζω ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε είναι να ορίσουμε ποιοι είναι οι βασικοί πολιτικοί γόρδιοι δεσμοί και γύρω από αυτού να μπορέσει το Κοινοβούλιο να επικυρώσει μια ισχυρή θέση. Εμείς κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συναπόφασης όπου μια κατακαιρματισμένη θέση του, του Κοινοβουλίου θα αποδυνάμωνε τη διαπραγματευτική μας θέση έναντι του Συμβουλίου. Το βασικό εμπόδιο είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Εμείς είχαμε άτυπες ανταλλαγές απόψεων στις συνεδρίασεις των συντονιστών αλλά αν πριν από το καλοκαίρι εμείς θέλουμε να συζητήσουμε τους βασικούς κανονισμούς Ιούνιο και Ιούλιο στην Επιτροπή Γεωργίας, αυτό απαιτεί ότι το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου θα παρουσιάσουμε τις εκθέσεις και θα τις παρουσιάσουμε στην μεταφραστική υπηρεσία. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι μέχρι τον Απρίλιο ή τα τέλη Απριλίου το Συμβούλιο θα μπορεί να έχει εγκρίνει μία θέση προς αυτή την κατεύθυνση. Φοβούμε λοιπόν ότι εγκρίνοντας εμείς μια θέση ως κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς ε, μία διαφορετική θέση από εκείνη του συμβιβασμού στο Συμβούλιο. Εγώ είχα τις πρώτες ανταλλαγές με την Δανή Υπουργό, της εξέφρασα τις επιθυμίες μας και επίσης ευχήθηκα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ε, μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ μας και επίσης το Συμβούλιο να να εγκρίνει ένα προσανατολιστικό έγγραφο είχα πει πριν από την Δανέζικη Προεδρία για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρύτερη βάση συζήτησης. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τη Δανέζα Υπουργό που θα έρθει αύριο και ελπίζω να επιμείνουν οι συνάδελφοι να έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς, άτυπους μηχανισμούς συνεργασίας με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλη αυτή την πορεία ε, αρμονικά. Θα είμαι σύντομος. Το πρώτο σημείο κλειδί γύρω από το οποίο θα πρέπει να ορίσουμε μία θέση του Κοινοβουλίου είναι η επανεξισορρόπηση της υποστήριξης εκ μέρους των κρατών μελών. Αυτό είναι και το πιο πολύπλοκο γιατί έχει να κάνει με την αναδιανομή των ε, <coughs> επιστροφών. Ξέρουμε ότι άλλες χώρες επιστρέφουν περισσότερο, άλλες λιγότερο. Οποιαδήποτε λοιπόν εξισορρόπηση θα, θα, ε, τον μεν θα οδηγούσε σε μία μείωση των ενισχύσεων για τους δε και υπήρξε ε, έντονη αντίσταση από τα κράτη-μέλη και αυτό γιατί φοβόντουσαν να χάσουν υποστήριξη στην ε, κοινωνία τους όπως επίσης ε, και πρόβλημα από τις χώρες οι οποίες θεωρούν ότι ακολουθώντας την κοινοτική νομοθεσία θα οπισθοδρομούσαν. Το ίδιο συμβαίνει και στο δεύτερο πυλώνα, όπου έχουμε μια διαφοροποιημένη κατανομή. Η Επιτροπή ενέκρινε μια διαφορετική προσέγγιση, χωρίς ε, να πειράζει την κατανομή του προπολογισμού. Και αυτές οι δύο πλευρές θα πρέπει να αξιολογηθούν από κοινού για να μπορέσουμε να καταλήξουμε χωρίς μεγάλες αλλαγές ε, στις ε, ενισχύσεις των κρατών μελών και να έχουμε δηλαδή μια πιο δίκαιη ισορροπία. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο ρυθμός σύγκλησης μέσα στα κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζουμε καλά σε πολλές ε, χώρες μέλη οι ενισχύσεις ε, κατανέμονται με διαφορετικούς τρόπους από περιφέρεια σε περιφέρεια με τεράστιες ανισότητες που δημιουργούν πολλά προβλήματα και πολλές φορές διακυβεύουν την ίδια την εθνική συνοχή. Θα πρέπει εμείς με αυτή τη μεταρρύθμιση να ορίσουμε έναν μηχανισμό σύγκλησης σύμβατο ε, για την εξέβριση ισορροπιών και μέσα στα κράτη-μέλη. Ένα άλλο σημείο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και γύρω από το οποίο θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες κατανόησης είναι το θέμα του greening, Όλοι συμφωνούν με το στόχο του greening, αλλά κανένας δεν συμφωνεί με τους στόχους ε, της Κομισιόν, με τις, τα λειτουργικά μέτρα της Κομισιόν για την προσέγγιση αυτού του στόχου. Εγώ θεωρώ ότι το greening θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο. Θα πρέπει να αποζημιώνει εκείνους τους γεωργούς οι οποίοι είναι πιο δυναμικοί ε, στο για το περιβάλλον. Όχι δηλαδή να τιμωρεί αυτούς που δεν δέχονται ορισμένες πρακτικές. Θα πρέπει εμείς ε, να μπορέσουμε να ε, αλλάξουμε τη θέση της Κομισιόν χωρίς όμως ε, να αποπροσανατολίσουμε το στόχο μας. Μια άλλη σημαντική πλευρά είναι ο ορισμός του ενεργού γεωργού όλοι συμφωνούν ότι θα, η τράπεζα θα πρέπει να είναι πιο επιλεκτική όταν επιλέγει τους δικαιούχους που θα πρέπει να είναι επαγγελματίες Γεωργή, ενώ η φόρμουλα που προτείνει η Κομισιόν δημιουργεί δυσκολίες και γύρω από αυτήν πρέπει να εργαστούμε. Για τις ε, πληρωμές ε, για τις συνδυασμένες πληρωμές. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και σε ορισμένες περιφέρειες η κατάργησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας με ό,τι θα, προέκυπτε από αυτό, όπως και το θέμα των δύο πυλώνων. Η Κομισιόν και εφιώς θα έλεγα θεωρεί το κάπινγκ ως ένα ε, μέσο για την χρηματοδότηση της καινοτομίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Η απόρριψη του κάπινγκ θα μπορούσε να διακυδέψει ένα μέρος των χρηματοδοτήσεων για την καινοτομία. Πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε πώς θα προσαρμόσουμε αυτόν τον μηχανισμό στους στόχους μας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, οι άμεσες πληρωμές, οι δορυφόροι και πάει που είναι όμως δευτερεύοντας, έστω και αν θα οδηγήσουν σε πολλές τροπολογίες και θα μας επιβάλλουν να καταλήξουμε σε μία προσέγγιση των θέσεών μας. Σε μία αρχική φάση πάντως εγώ προτείνω να συγκεντρωθούμε γύρω από αυτά τα 5-6 σημεία κλειδιά τα οποία είναι ουσιώδη από πολιτικής πλευράς για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μία ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου. Είμαι στη διάθεσή σας ε, για τη συνεργασία που θα μας οδηγήσει να βρούμε λύσεις όσο το δυνατόν πιο συμμερισμένες από την πλειοψηφία για να μπορέσουν να αντιπαρατεθούν στο Συμβούλιο και να, να αντιμετωπίσουν την αξιολόγηση της Κομισιόν. Έχω και άλλες παρατηρήσεις να κάνω, οι οποίες δεν είναι όμως πια τόσο σημαντικές αυτή τη φάση. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο και περιμένω τις θέσεις σας. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε όπως και τους αντιπροέδρους ε, για την εκλογή σας. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε την εξαιρετική εργασία που κάναμε στην πρώτη, στο πρώτο τμήμα της θητείας. Ευχαριστώ Λουίς. Βλέπω ότι έγινε πολύ καλή δουλειά. Ξεκινάει η συζήτηση. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να κρατήσουν το χρόνο τους, να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσει να μιλήσει και ο Μισελ Νταντά. Ο κύριος Βαγεσόφσκι και μετά ο Μάρτιν Όσλιν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα σας συγχαρώ και εγώ και θα εκφράσω την πεποίθησή μου ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Μία ερώτηση προς τον εισηγητή. Στο, στη μελλοντική εργασία μας προβλέπεται να κάνουμε αναλύσεις εμπειρογνωμόνων για τις απευθείας πληρωμές για να δούμε εάν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συνθήκης. Έχουν προκληθεί ορισμένε αμφιβολίες σχετικά με αυτό το ε, λεγόμενο greening διότι στη συνθήκη το greening, η περιβαλλοντική προστασία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν περιλαμβάνεται λοιπόν στη, στους ε, αντικειμενικούς σκοπούς της ε, ΚΑΠ ε, στα πλαίσια της συνθήκης. Δεν θα πω βέβαια σε λεπτομέρειες οι σκοποί που περιλαμβάνονται στο κείμενο είναι διαφορετικοί και επαναλαμβάνω το greening απουσιάζει από τις διατάξεις της συνθήκης. Το ίδιο πρόβλημα ανακύπτει σχετικά με την κατανομή πληρωμών μεταξύ χωρών μελών. Στο άρθρο 18 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχει ρητή απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος ουδήποτε λόγω εθνικότητας. Όμως, ιστορικά, οι πληρωμές γίνονται όχι με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά με βάση την εθνικότητα των αγροτών. Και αυτό νομίζω αντιβαίνει στο 18 της συνθήκης. Στο δε άρθρο 39 βρίσκομαι διατάξεις σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα αντικειμενικά κριτήρια. Και εκεί αναφέρονται περιφερειακέ ιδιαιτερότητε, οι περιφερειακές διαφορές, όχι όμω περιφε... όχι όμως εθνικές διαφορές. Και υπάρχει και το άρθρο 40, το οποίο απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση σε βάρο αγροτών τη ενώσεω. Κατά την άποψή μου, τα διαφορετικά επίπεδα πληρωμών είναι αποτέλεσμα διακρίσεων και αυτό πρέπει να αναλυθεί και νομικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να παραπέμψουμε το θέμα στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή τι γνώμη έχει για την πρόταση μου αυτή. Ο Μάρτιν Χόσλινγκ και μετά η κυρία Μαγκίνες. Ο Μάρτιν. Και από τη δική μας πλευρά συγχαρητήρια ε, για την εκλογή του νέου Προεδρίου ή του παλαιού τέλο πάντων όπως θέλετε το βλέπετε. Εγώ περίμενα σήμερα ο εισηγητής να υποβάλει κάποιες νέες προτάσεις και ιδέες. Διότι ασκείται κριτική στις προτάσεις, αλλά και το Κοινοβούλιο μάλλον έχει περιοριστεί σε κριτική και όχι σε υποβολή δικών του προτάσεων. Ας μην περιμένουμε λοιπόν πολύ μέχρι να καταθέσουμε νέες ιδέες και προτάσεις. Και δυστυχώς κύριε Σιγητά, Σήμερα δεν είδα διόλου να το κάνετε αυτό. Ότι οι Υπουργοί Γεωργίας προφανώς δεν είναι σε θέση να κάνουν προτάσεις διότι όλοι σκοτώνονται μόνο για την κατανομή των πόρων, αυτό δεν μας εκπλήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει εκείνο να καταθέσει πρωτοβουλίες και προτάσεις. Και αυτό που είπατε τώρα για την κατανομή μεταξύ των χωρών μελών, η πρόταση στο σημείο αυτό είναι ανεπαρκής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη κατανομή πληρωμών εντός τη ενώσεως. Δεν αρκεί ωστόσο μόνο να διαπιστώνουμε τις αδικίες. Εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα αυτή που δεν βλέπουν από το εθνικό επίπεδο. Από το δεύτερο πυλώνα οι νέε χώρε μέλη έχουν περισσότερα χρήματα, αλλά πολλές χώρες δεν μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν πλέον τις δαπάνες του δεύτερου πυλώνα. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αντιστάθμιση. Για δε το πρασίνισμα, το greening, βρίσκω ότι η πρόταση σχετικά με τις συστημικές κατατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί αντικειμενικά. Αλλά γιατί άραγε δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε όλα αυτά εθελοντικά κατάλαβα από αυτά που είπε ο κύριος Καπούλα Σάντος ότι ίσως να γίνει προσφορά ή οικειοθέλης, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Οι στόχοι του πρασινίσματος πρέπει να είναι δεσμευτικοί. Η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα πρέπει επίσης να περιληφθεί στους στόχους, γιατί είναι κεντρικό θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και το ίδιο για την κλιματική αλλαγή, η προστασία δηλαδή. Δεν μπορούμε να βάλουμε κατ' επιλογή ορισμένα ζητήματα. Εμάς βέβαια δεν μας αρέσουν οι προτάσεις. Δεν ξέρω για παράδειγμα για το ποσοστό του 70% στους χυμούς εάν είναι πραγματικά σωστό. Για τα 7% που αναφέρατε προηγουμένως για μέτρα περιμένω να δούμε να μας πούν ακριβώς τι θα πούν για ζώνες προστασίας των ε, νερών ή προστασία ορισμένων τμήματων των ε, γεών κλπ. Αλλά αυτά πάντως είναι νούμερα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και που δεν μπορούμε βέβαια να τα μειώσουμε ιδιαίτερα. Το ερώτημα ποιος είναι αγρότης μου φαίνεται και αυτό σωστό να συζητηθεί. Γιατί η κατανομή των πληρωμών αλλά και σχετική αιτιολόγηση θα πρέπει να απευθύνεται στους σωστούς παραλήπτες και υπάρχει πρόβλημα βεβαίως. Υπάρχουν οι εκμεταλλεύσεις που δεν χρειάζονται καν υποστήριξη. Το 5% πρέπει να προέρθει από τη Γεωργία, σύμφωνα με την πρόταση. Είναι δύσκολο, το βλέπω και εγώ, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα καταγράψει όλα. Πάλι όμως και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Και ναι, είναι επικίνδυνη η γραφειοκρατία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να καταθέσουμε στο αρχείο τα θέματα. Για τον περιορισμό, εμείς είπαμε πάντοτε ότι πρέπει να αρχίζουμε στα 150.000 και οι 300.000 δεν είναι θέμα για τις 99% των εκμεταλλεύσεων στην Ένωση. Και η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι τρομερά υπερβολική. Στη Γερμανία ίσως αναφέρεται σε 4 ή 5 δωδεκάδες εκμεταλλεύσεων Άρα ο περιορισμός πρέπει να αρχίζει, ο ορισμός δηλαδή νωρίτερα και σταδιακά να αρχίζει δηλαδή κάτω από τις 100.000 ώστε να δώσει και πραγματικά κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί 300.000 πληρωμών αν βάλει κανείς μέσα και και τα εργατικά χέρια δεν μπορεί να αναφέρεται παρά μόνο σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν αποκαθιστά δικαιοσύνη. Και ένα τελευταίο, θα το τονίζουμε σε κάθε συνεδρία γιατί βλέπουμε να λείπει εδώ. Σήμερα η Γερμανική Ομοσπονδία Αγροτών ζητάει ειδική στρατηγική για το Λεύκομα και οι αγρότες γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος από το 80% εξάρτησής μας από εισαγωγές λευκόματος και αν δεν κάνουν προτάσεις άλλοι θα πρέπει να τις κάνουμε εμείς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό για τη μελλοντική μεταρρύθμιση. Η κυρία Μαγκίνες και μετά η κυρία Γέγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κάπουλα Σάντος ε, για την παρουσίασή σας. Θα συμφωνούσα με τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι να διαμορφώσει κανείς πραγματικές αναρακτικές προτάσεις. Όσο δύσκολο όμως και αν είναι, εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό και να βρούμε τομείς κλειδιά που θέλουμε να αλλάξουμε και όπου θέλουμε να συμβάλλουμε θετικά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μπλέξουμε σε λεπτομέρειες τη συζήτηση και αυτό θα ήταν λάθος. Θα ήθελα λοιπόν να ε, εντοπίσουμε ε, έξι ε, σημαντικούς τομείς στο θέμα των άμεσων ενισχύσεων στο οποίο όπου μπορούμε πραγματικά να κάνουμε κάτι. Να ξεκινήσω από το πρασίνισμα, από τις το να είναι φιλική προ το περιβάλλον η Γεωργία. Ε, στην αρχή το Κοινοβούλιο μα είχε κάποιε πολύ καλέ ιδέε ε, για ε, το πρασίνισμα αυτό και δυσαρεστήθηκα που είδα ότι η Κομισιόν έχει περιορίσει τον ορισμό του πρασινίσματο σε τρει συγκεκριμένου τομεί. Θα τροποποιήσουμε λοιπόν την πρόταση για να προσπαθήσουμε να σωματώσουμε αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο από την αρχή. Ίσως να είναι δύσκολο για την ε, Κομισιόν ε, όσον αφορά τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με ε, την Κομισιόν και να υποβάλουμε κάποιες επικοδομητικές ιδέες ώστε να επιτρέψουμε την καινοτομία, να, να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις όσον αφορά το νερό και ήδη έχουμε στηρίξει αυτήν την την ιδέα, αλλά έχουμε μια πιο ευρία, ε, ένα πιο ευρύ όραμα όσον αφορά το πρασίνισμα. Ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό, αλλά δύο θέματα που αφορούν το greening είναι το ένα, το 30%, η κατανομή του 30%. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι το ποσοστό αυτό είναι υπερβολικά υψηλό, άλλοι ότι είναι πολύ χαμηλό θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Νομίζω όμως ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ε, ένα τμήμα των άμεσων ενισχύσεων που συνδέεται με, μέσα, μέτρα περιβαλλοντικά και κλιματικά και θα πρέπει να καθορίσουμε ε, πού ακριβώς στοχεύει το μέτρο αυτό. Έχω μια ανησυχία όσον αφορά τι πράξει κατεξουδότηση, όσον αφορά το πρασίνισμα και άλλα μέρη τη πρόταση αυτή. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα συνεργαστεί μαζί μα ώστε να κατανοήσουμε απόλυτα τι συνέπειες του να επιτρέψουμε ε, τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση όπως προτείνονται. Ε, χρειάζεται όμω να γίνει ει βάθος ανάλυση όσον αφορά τι συνέπειες. Να ε, προχωρήσω σε κάποια πιο γενικά θέματα όσον αφορά το θέμα του προπολογισμού και την κατανομή του στα κράτη-μέλη. Το θέμα αυτό είναι πολιτικά πολύ ευαίσθητο και για μας και για το Συμβούλιο. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα αυξάναμε τον προπολογισμό και όλοι θα είχαμε πιο υψηλά επίπεδα. Στον πραγματικό κόσμο όμως ε, μοιράζουμε ένα μικρότερο ποσό σε περισσότερα και θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν μιλήσαμε για ισότητα ούτε για αμεσότητα και κάποια κράτη-μέλη ανησυχούν ε, σχετικά με τις ανισότητες. Ε, δεν γνωρίζουμε το ακριβώς μέγεθος του προϋπολογισμού. Ε, θα πρέπει όμως πολιτικά να είμαστε κουρτισμένοι εντό εισαγωγικών και να αναγνωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αν πρόκειτο να ανακατανύμουμε ίσα σε όλα τα κράτη-μέλη θα υπήρχαν σημαντικές συνέπειες, αρνητικές για πολλά κράτη-μέλη και κάτι τέτοιο μπορεί πολιτικά να μην γινόταν αποδεκτό. Γι' αυτό ξεκινάμε με αυτή την προοπτική. Είχα διάφορες συζητήσεις και ξέρω ότι τα παλαιά και τα νέα κράτη-μέλη είχαν αναλυτικές ε, συζητήσεις σχετικά με τις ανησυχίες τους. Είχα και συναδέρφους από τα παλαιότερα κράτη-μέλη που ανησυχούσαν ε, όσον αφορά την ανακατανομή μεταξύ των παλαιών κρατών μελών και θα πρέπει να εξεταστεί αυτό αυτό. Συμπεριλαμβάνου του θέματος, ε, συμπεριλαμβανομένου του θέματος εάν θα συμπεριλάβουμε όλον τον προπολογισμό, τον ε, πυλώνα 1 και 2. Υπάρχουν όμως ακόμα, ε, ε, είναι ακόμα αβέβαιος ο προϋπολογισμός, θα συναντήσουμε λοιπόν δυσκολίε ε, κατά την εξέβρεση συμφωνία εντό τη Επιτροπή μα ε, για την ε, κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Παρόμοια δυσκολία υπάρχει όσον αφορά την κατανομή στου γεωργού εντό του, του κάθε κράτου μέλου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάποια κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο μετάβαση από τι περιφερειακέ πληρωμέ θα δεχτούμε το χρονοδιάγραμμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι υπερβολικά ε, γρήγορη η αλλαγή αυτή για κάποια κράτη-μέλη και θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχει κάποιο βαθμό ευελιξία για να μην διαταράξουμε την παραγωγή και τη γεωργία εντό των κρατών μελών, αποδεχόμενοι ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ. Αυτή είναι η δυσκολία που συναντάμε. Κατά τη γνώμη μου, αυτέ είναι οι πιο πολύπλοκε μεταρρυθμίσει ε, που είδαμε ποτέ και που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ε, πολιτικοί. Διότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα πληρωμών και διάφορες συνθήκες και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις διαφορές και να ε, εργαστούμε προς την εξέβρεση λύσης. Ε, ταυτόχρονα θα ήθελα να αμφισβητήσω αν είναι δυνατόν να, φτάσουμε στην ενιαία αξία αυτή μέχρι το 2019 σύμφωνα με τον ισχυρισμό. Νομίζω ότι είναι πολύ σφιχτό αυτό το χρονοδιάγραμμα ε, μάλλον δεν είναι ούτε ρεαλιστικό ούτε ε, πραγματοποιήσιμο. Έχω μια ευρύτερη ερώτηση προς την Κομισιόν. Τι όραμα έχει, ε, ποια είναι η λογική του να συνδέσουμε τις πληρωμές με τις εκτάσεις για την μακροπρόθεσμη επιβίωση τη κοινή γεωργική πολιτική. Ε, σήμερα γιορτάζουμε τα 50 χρόνια τη κοινή γεωργική πολιτική. Αν διαβάσετε τι έρευνε ε, σχετικά με τη ε, διασύνδεση των ενισχύσεων με, το, με τι εκτάσει, αυτό δεν είναι ο ιδανικό τρόπο να στηρίξουμε την γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν μακροπρόθεσμε συνέπειε μια τέτοια εξέλιξη. Όσον αφορά τον ορισμό του ενεργού γεωργού, η Κομισιόν ήταν πολύ σαφή στο θέμα αυτό και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω των ε, επιφυλάξεων που εξέφρασε το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι αρκετά σαφές. Εμεί θέλουμε έναν ορισμό ο οποίος να είναι φιλικός προς τον χρήστη, για τα κράτη-μέλη δηλαδή και για τους γεωργούς. Για του περισσότερου γεωργού, ε, προφανώ ε, αυτό δεν είναι θέμα, διότι γνωρίζουν ότι είναι ενεργοί, αλλά ο νομικό ορισμό ε, θα είναι πολύ σημαντικό, διότι είτε θα μπορεί να εφαρμοστεί πολύ εύκολα, είτε θα είναι πολύ πολύπλοκη η εφαρμογή του ορισμού αυτού. Και εξάτασα τρόπους αλλαγή του συστήματος θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι καλύτερα σε θέση να κρίνουν ποιος είναι ενεργός γεωργός και ποιος όχι. Γνωρίζω όμως ότι από το ελεγκτικό συνέδριο ότι αυτό θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε έναν ορισμό. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε γεωργό θεωρεί ότι ο γείτονα δεν είναι εξίσου ενεργό με αυτόν. Ε, θα πρέπει να πετύχουμε μια συμφωνία με του γεωργού για το θέμα αυτό. Εάν όμω δεν ε, βρούμε καλύτερο ορισμό, θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον παλιό. Όσον αφορά την πρόβλεψη ανώτατου ορίου, το κάπινγκ. Το κάπινγκ δεν συμπεριλαμβάνει το πρασίνισμα. Το πρασινίσμα ε, εξαιρείται από το κάπινγκ, από την πρόβλεψη ανώτατου ορίου ε, και αυτό λοιπόν αποτελεί πολύ ενδιαφέρον ε, μέρος της πρότασης. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη για το κάπινγκ. Κάποιοι συνάδελφοι όμως λόγω των δομών στα κράτη-μέλη τους έχουν απόψεις και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε συμβιβασμό όσον αφορά την πρόταση αυτή. Για άλλα κράτη-μέλη δεν αποτελεί πρόβλημα. Όσον αφορά ε, τα δικαιώματα, διαπίστωση των δικαιωμάτων, ε, Έχουμε εδώ το έτος 2014 σε σχέση με το 2011. Ε, πιστεύω και πάλι ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρει μία μέθοδο πιο φιλική προς τον Γεωργό, όπου να μην συνδέουμε το θέμα αυτό των δικαιωμάτων με τρόπο που να δημιουργήσει περιττές αντιδράσεις ε, από τους γεωργούς όσον αφορά ε, την ε, μίσθωση γεών. Ίσως και εδώ η Κομισιόν να μπορεί να βρει τρόπο να βρεθεί ευελιξία πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τους ίδιους στόχους. Κάποιε λεπτομέρειε Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Όσον αφορά τους νέους γεωργού. ε, χρειαζόμαστε μια ε, πρακτική λύση. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από απλά να μιλάμε για αυτού. Ε, όλοι είναι υπέρ των νέων γεωργών, όπως όλοι είναι υπέρ των γυναικών ε, στην πολιτική, αλλά πολύ λίγες δράσει αναλαμβάνονται που ε, πετυχαίνουν αλλαγή της κατάστασης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η στήριξη που δίδεται έτσι στους νέους γεωργούς ουσιαστικά δεν πετυχαίνει τίποτε. Αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε κάτι θα πρέπει να εξετάσουμε το μέτρο αυτό και να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα για τους νέους γεωργούς, διότι αυτή είναι το μέλλον μας. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Έχω και κάποιες άλλες ε, λεπτομέρειες, αλλά το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω εδώ, διότι θα το ξανασυζητήσουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με τους μικρούς γεωργούς. Όπως ε, μου είπε ένας συνάδελφος, ε, είναι θέμα μικρών δικαιούχων. Θα πρέπει να εξετάσουμε πόσα κράτη-μέλη θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το μέτρο και ποιε θα είναι οι συνέπειες ενό τέτοιου προγράμματο. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα που αφορούν τον πυλώνα 2 ε, σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Γενικά, οι παρατηρήσει μου για τις άμεσες ενισχύσει είναι ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό για τους γεωργούς στα κράτη-μέλη. Το μόνο που θα μας ρωτήσουν είναι τι συνέπειε θα έχει αυτό στι πληρωμέ που λαμβάνω εγώ, διότι αυτό θα επηρεάσει τον προγραμματισμό του και πραγματικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε για κάθε άτομο ε, τι συνέπειε. Θα πρέπει όμω να του πείσουμε ότι ό,τι και να κάνουμε δεν θα οδηγήσει σε ε, ε, δραματικές ριζικές αλλαγέ προ το χειρότερο. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν χρόνο να προσαρμοστούν και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα νέο καθεστώ θα είναι καλά σχεδιασμένο, διότι έχω την ανησυχία ότι ακόμα και αν πετύχουμε όλους τους στόχους μας με εκθέσεις, τροπολογίες και διαπραγματεύσεις, Ακόμα και αν πετύχουμε δηλαδή ένα νέο ε, σύστημα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, είναι πολύ σφιχτό αυτό το χρονοδιάγραμμα και πιθανότατα κάτι τέτοιο να μην είναι εφικτό. Ε, αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου προς τον εισηγητή. Τον ευχαριστώ για τη δουλειά που έχει κάνει. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά και εγώ με προσοχή θα ακούσω τους συναδέρφους ώστε να προσπαθήσω ε, να λάβω υπόψη μου τις ανησυχίες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάιραντ. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γέγελ και μετά ο Τζορτζ Λάιον. Ευχαριστώ. Και από τη δική μου πλευρά Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Όλοι αναμένουμε βεβαίως να συνεχιστεί η αγαστή μας συνεργασία. Αυτό, αυτή η πρώτη έκθεση για τις άμεσες πληρωμές δείχνει που το το Σε Ευχαριστώ τον κύριο Κάπουλος, Κάπουλα Σάντος για τα λόγια του. Βέβαια ελπίζω ότι θα συγκεκριμενοποιηθούν τα όσα προτείνει και ελπίζω στο προσεχές μέλλον όταν λοιπόν θα φέρει συγκεκριμένε προτάσει, τότε θα τις συζητήσουμε ξανά. Έχοντα παρακολουθήσει τα όσα είπαν οι άλλοι συνάδελφοι, θέλω να σημειώσω δύο θέματα που νομίζω ότι είναι αμφιλεγόμενα. Βέβαια θα χρειαστεί να καταλήξουμε σε κάποια λύση, αλλά και ε, να μην λησμονούμε ότι ως Γερική Επιτροπή δεν είμαστε και ο ομφαλός της γης. Άλλες πέντε επιτροπές, έξι συνολικά, ασχολούνται με το θέμα αυτό και καλά θα κάνουμε να συνεργαστούμε μαζί τους και να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις. Η δεν θα επιτύχουμε. Αυτό το πρώτο σχόλιο μου. Το δεύτερο, οι άμεσες αυτές πληρωμές, αλλά και ολόκληρη συζήτηση που στρέφεται γύρω από αυτές, δείχνει σε όλες και όλους μας, στις συζητήσεις δηλαδή, στις χώρες μέλη, με τους αγρότες και με τους πολίτες, μας δείχνουν και πού βρίσκονται οι ευθύνες για τη διαχείριση των χρημάτων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και πόσα θα λάβουμε αλλά και πώς θα πορευτούμε μέχρι ό,τι τα λάβουμε ως Γεωργική Επιτροπή και τελικά πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, πόσα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με καλές προτάσεις ή μη θα ιτηθούμε στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο του προπολογισμού για τη Γεωργία. Προσωπικά βλέπω δύο πραγματικά προβληματικά σημεία Πρώτον, τον ενεργό αγρότη. Όλοι θελήσαμε να υπάρξει μια καλύτερη διατύπωση, μια καλύτερη περιγραφή του τι σημαίνει ενεργός αγρότης. Αλλά αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγουν πολλές δυνατότητες για διαφορετικές ερμηνείες και δεν εξυπηρετεί. Δεν μπορεί να θέλουμε μεγάλες εκμεταλλεύσεις να εισέλθουν στην γεωργία και να μπορούν να απορροφούν όσα αγροτικά κονδύλια θέλουν. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι γεωργοί είτε ε, είναι κατά κύριο επάγγελμα είτε κατά δευτερεύουσα δραστηριότητα γεωργοί να μπορούν να ζήσουν τη δραστηριότητα τους αυτή. Και το επόμενο είναι το πρασίνισμα, το greening. Έχω πει κατά επανάληψη ότι δέχομαι κατά 100% την πρόταση να γίνει δεσμευτική στον πρώτο πυλώνα η greening. Γιατί το δεύτερο πυλώνα δεν εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά. Χρειαζόμαστε όμως και για την αποδοχή της CAP. Και ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Τώρα το πώς θα διαμορφωθεί το πρασίνισμα αυτό νομίζω αυτό θα οδηγήσει και σε άλλες πολλές συζητήσεις. Το γεγονός τώρα ότι οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις απελευθερώνονται από ελέγχους εξαιρούνται από ελέγχους. Κάτι τέτοιο δεν μπορώ να δεχθώ, ούτε πρόκειται να το δεχθώ. Ούτε άλλωστε θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Εδώ δεν επιτρέπεται να κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός. Και οι παραδοσιακοί γεωργοί δρούν σύμφωνα με τις ορθές παραδοσιακές πρακτικές και αυτό οφείλει να τιμηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ελίζαμπεθ ο George Λάιον και μετά ο κύριος Κόσιντζερ. Ευχαριστώ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοί μου. Σας συγχαίρω και πάλι και εσάς ως πρόεδρο και τους αντιπρόεδρους. Θα είμαι σύντομος, θα περιοριστώ σε σημαντικά θέματα. Υποστηρίζω το πλαίσιο που έχει καθορίσει η Επιτροπή για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Άλλωστε θα ήταν παράξενο να αντιταχθούμε διότι λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις σε μεγάλο βαθμό που έχουν περιληφθεί στις δύο εγκεκριμένε από το Κοινοβούλιο εκθέσεις και στην προηγούμενη δηλαδή έκθεση την οποία είχα την τύχη να συντάξω. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία για το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειε. το πρώτο θέμα είναι πρέπει να δούμε ποια μορφή λαμβάνει η νέα ΚΑΠ, αλλά αυτό είναι δύσκολο διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εκτελέσει πολλά μέσω εκτελεστικών πράξεων και καταξιδότηση πράξεων. Πρώτος στόχος του Κοινοβουλίου θα, έπρεπε να, θα πρέπει να είναι να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει περισσότερο τι προτίθεται να κάνει με τη χρήση των οργάνων αυτών, των πράξεων αυτών και όχι να τα χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε ελευθερία ίδια επιλέξει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Το δεύτερο που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε νομική γνωμοδότηση για το ποιο ρόλο η παρούσα επιτροπή μας σχετικά με την κατανομή των πληρωμών μεταξύ των χωρών μελών, που είναι θέμα κλειδί και που επαναλαμβάνεται σε κάθε συζήτηση που διεξάγουμε. Και όταν συζητούμε με το γραφείο του Επιτρόπου, αλλά και με τους κοιόδης συγητές, το, τα μέλη του γραφείου του Επιτρόπου μας είπαν καθαρά ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αλλάξουμε τα, τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων είναι μέσω των παραρτημάτων, γιατί οι νέοι κανονισμοί προβλέπονται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς λέμε ότι ο μόνος μηχανισμός που έχουμε είναι να τροποποιήσουμε τα ποσά του πίνακα στο τέλος του παραρτήματος. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να συζητηθούν στην Επιτροπή μας. Θα προτείνω λοιπόν στον Πρόεδρο και στον εισηγητή να ζητήσουμε νομική γνωμοδότηση σχετικά με το ποιε αρμοδιότητες έχει η Επιτροπή μας αλλά και το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων. Γιατί η απάντηση φοβούμαι ότι θα είναι πολύ μικρέ δυνατότητες έχετε διότι περιλαμβάνονται τα ποσά αυτά στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ίσως λοιπόν, εάν το γνωρίζουμε αυτό, να αποφύγουμε μάταιες πολιτικές προσπάθειες και κινητοποίηση. Εάν είναι μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, Αυτό περιορίζει τη δυναρμοδιότητα του Κοινοβουλίου στο να πει μονάχα ναι ή όχι. Και άρα η επιρροή που μπορεί να ασκήσει το Κοινοβουλίο μειώνεται. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, να μα απαντήσει δηλαδή στην ερώτηση ποιε συγκεκριμένε εξουσίε έχουμε σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού της ΚΑΠ για το πολύ συγκεκριμένο αυτό και σημαντικό θέμα. Πολύ σύντομα τώρα ορισμένα άλλα για τις βασικές άμεσες πληρωμές υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την περίοδο προσαρμογής, αν δηλαδή το 2019 επαρκεί για τις χώρες μέλη για να κάνουν αυτές τις προσαρμογές, αλλά και το έτος αναφοράς των ε, απαιτήσεων του 2011 δηλαδή για το νέο καθεστώς. Υπάρχει πάλι ένα ερώτημα εδώ σχετικά οι γεωργοί, εάν κάνουν τις αιτήσει τους με βάση το 2011, πώς θα μπουν στο νέο πλαίσιο, εάν δεν έχουν κάνει, μάλλον, τις ε, αιτήσει του 2011. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως αυτό το 2011 ως έτος αναφοράς και μόνο του είναι πολύ περιοριστικό. Υπάρχουν και δύο άλλα σημαντικά θέματα. Η οροφή και ο ενεργός αγρότης. Αρχίσαμε να τα συζητούμε αυτά και βλέπουμε τώρα τις απαιτήσει για τον ενεργό αγρότη που θα πρέπει να μπορεί στις 15 Μαΐου να δηλώσει ότι το συνολικό το αγροτικό ε, εισόδημα δεν είναι λιγότερο του 5% του συνολικού του εισοδήματο. Και αυτό ε, δεν μπορεί να γίνει παρά δύο χρόνια μετά που θα είναι ε, ε, συμπληρωμένα τα βιβλία του. Εγώ βρίσκω το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και πολλοί που θα θεωρήσουν ότι τη δυσκολία την προκαλεί το πρασίνισμα θα αρχίσουν να ρωτούν θέματα σχετικά ποιος είναι ο εργαζόμενος στη γεωργική εκμετάλλευση, αν χρειάζεται ε, η τήρηση βιβλίων και με ποιους κανόνες και αυτά όλα είναι περιπλοκότητα που θα κοστίσουν στις χώρες μέλη, θα είναι δαπανηρές για τις χώρες μέλη αυτά τα δύο μέτρα. Για το πρασίνισμα συμφωνώ και με τα όσα είπαν άλλοι πριν από μένα. Πρώτον ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο το, πρόγραμμα και δεύτερον ότι δεν είναι αρκετά εύκαμπτο για να μπορεί να λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες πολλών χωρών μελών. Μου φαίνονται τα μέτρα αυτά ότι είναι κάπου ενία για όλες τις χώρες. Και το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να είναι και δεσμευτικά, υποχρεωτικά για όλους τους γεωργούς ή θα είναι υποχρεωτικό για τις χώρες μέλη να προσφέρουν δυνατότητα στους γεωργούς και αυτοί θα αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι ένα σύστημα κινήτρων είναι πολύ καλύτερο και λειτουργεί καλύτερα για να ε, δώσει τη δυνατότητα στους γεωργούς να κάνουν και τη λεγόμενη cross-compliance. Για τους νεαρούς γεωργούς συμφωνώ με την αρχή. Η πρόταση είναι καλή. καθώς και η δυνατότητα διατήρησης των συνδεμένων πληρωμών. Με αυτά τα λίγα σχόλια λοιπόν Πρόεδρε Ελπίζω να έχουμε θετικές απαντήσεις του εισηγητή, γιατί όπως είπα χρειαζόμαστε ασφάλεια σχετικά με, το, με την κατανομή των άμεσων πληρωμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ζόρζο. Ε, θα δώσω το λόγο στον Κώστιγκερ. Αλλά πρέπει να σου πω όμως ότι εμείς δεν έχουμε κανέναν περιορισμό επισήμως μπορούμε να αλλάξουμε και τον χρηματοδοτικό πίνακα και μετά πρέπει να το ψηφίσουμε φυσικά. Αυτό θα, αυτή η αλλαγή θα δημιουργούσε πρόβλημα τόσο στο Συμβούλιο όσο και σε εμά. Οπότε μπορούμε να, πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, αλλά επίσημα μπορούμε εμείς να τροποποιήσουμε όλες τις προτάσεις της Κομισιόν και τους χρηματοπι... χρηματικούς πίνακες. Κυρία Κώστιγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για τις ε, πρώτες ιδέες του και τους συλλογισμούς που μας παρουσίασε. Συμμερισώ με τη θέση του ότι υπάρχουν εδώ ε, κάποια σημεία που θα πρέπει να συζητήσουμε και η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να υποβάλει ε, συγκεκριμένες προτάσεις ε, και εναλλακτικέ λύσεις ώστε να διασφαλίσουμε το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη. Συμφωνώ ότι τα μέτρα για το πρασίνισμα που προτείνονται είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να πετύχουμε ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε και ποιος είναι ο προϋπολογισμός ε, και πιστεύω ότι ε, οι στόχοι ότι τα μέτρα που αναφέρονται εδώ πέρα δεν συνάδουν με τους στόχους μας. Πιστεύω ότι είναι λάθος ε, δρόμος, διότι ε, νομίζω ότι η μείωση της παραγωγής αυτή τη στιγμή αντίκειται στους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ε, είναι επίσης... Η πείρα μας μας δείχνει ότι ε, τα θέματα αυτά προκαλούν πολύ έντονες συζητήσεις μεταξύ των γεωργών που δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ε, δεν μπορούν να καλλιεργούν μέρος των εκτάσεών τους. Τα τελευταία χρόνια ε, έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για χαρτογράφηση των εκτάσεων. Όλα αυτά μάταια έγιναν. Νομίζω ότι πολλοί ε, δεν θα μας καταλάβουν και αυτό δεν βοηθάει και στην αποδοχή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επίσης θα ήθελα να ε, επιστήσω την προσοχή σας ε, στο γεγονός ότι αν τα κάνουμε αυτά, στο μέλλον θα πρέπει να διεξάγουμε και την συζήτηση γιατί οι γεωργοί λαμβάνουν πληρωμές για να μην καλλιεργούν εκτάσεις για την αγρανάπαυση. Θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή και Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να καθοδηγούμαστε και από τις συζητήσεις που γίνονται από το κοινό. Πάντως θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους ότι ε, ότι και όσον αφορά τον ε, προϋπολογισμό και εδώ η αγρανάπαυση ουσιαστικά αντίκειται σε αυτά που ψηφίσαμε πριν κάποιους μήνες η Ευρώπη θα πρέπει πραγματικά να σκεφτεί πώς μπορεί να ε, κλείσει το κενό αυτό ε, στην πρωτεΐνη, στη διατροφή. Και την, την έλλειψη ε, λευκόματος που θα υπάρχει στο, στο μέλλον στη διατροφή και δεν ξέρω σε τι βαθμό οι συνάδελφοι γνωρίζουν τα δημοσιεύματα των τελευταίων ε, ημερών ε, και αυτά που έχει πει το Ελεκτικό Συνέδριο που ε, επικρίνει έντονα τις προτάσεις της Κομισιόν και που θεωρεί ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής με τα προτινόμενα μέτρα. οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας ε, σίγουρα θα οδηγήσουν σε αύξηση της γραφειοκρατίας και κάποιος που ασχολείται εδώ και αρκετό καιρό με την ε, γεωργική πολιτική θα το γνωρίζει αυτό. Ε, θα έχουμε περισσότερους ελέγχους, περισσότερη γραφειοκρατία και αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό πρόβλημα. Ο Επίτροπο, στα πλαίσια της πράσινη Εβδομάδας ε, ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη μόνα τους ε, δημιουργούν αυτή την ε, γραφειοκρατία. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινεί. και να εξετάσουμε ποια κράτη-μέλη έχουν το μικρότερο περιθώριο λάθους και είναι αυτά που έχουν τους πιο συχνούς ελέγχους και και θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να διασφαλίσει τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Ε, κάτι τέτοιο δεν είναι απλό. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι θα πρέπει να δούμε μαζί τους δύο πυλώνες της κοινή γεωργικής πολιτικής και να μην τους συστήσουμε ξεχωριστά τον έναν από τον άλλον η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι κεντρικό σημείο της κοινή γεωργικής πολιτικής σε πολλά κράτη-μέλη και ελπίζω σύντομα να λάβουμε απαντήσεις ε, στο τι θα κάνουμε σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη ήδη έχουν δημιουργήσει πολύ καλή πολιτική τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν και την υποδοχή, αποδοχή των, ε, των γεωργών ε, τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση αυτών των κρατών μελών που λόγω του πρασινίσματο ε, θα πρέπει ε, να κάνουν περικοπές στα προγράμματα αυτά. Πώς μπορούμε να βρούμε λύσει, ε, διότι νομίζω ότι το χειρότερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε στους γεωργούς μας είναι να καταργήσουμε υπάρχοντα επιτυχή προγράμματα με μια μεταρρύθμιση η οποία δεν είναι απαραίτητη. Θα πρέπει όλοι όσο γίνεται πιο γρήγορα να βρούμε εναλλακτικέ ε, λύσεις ώστε τα επιτυχή υπάρχοντα προγράμματα που πάνε στα κράτη-μέλη να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ε, είναι πολύ σημαντικό το σύστημα των ε, κινήτρων και το κράτος μέλος μου. Η η πατρίδα μου δείχνει ότι το σύστημα κινήτρων αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε, διότι ε, στην χώρα μου υπάρχει μεγάλη αποδοχή ε, της ε, γεωργικής πολιτικής από τους γεωργούς. Επανειλημμένα, έχει αναφερθεί ότι θα πρέπει να πετύχουμε την αποδοχή των καταναλωτών και των φορολογουμένων. Νομίζω ότι και στους γεωργούς θα πρέπει να πετύχουμε το ίδιο πράγμα, που εργάζονται σκληρά ώστε να διασφαλίσουν την, ε, ε, την ε, τροφοδοσία της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να λάβουμε υπόψη μας τους ανθρώπους απέναντι στους οποίους λογοδοτούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιξ και μετά ο Σέρτζο Σιλβέστρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέλφους που ήδη μίλησαν. Στην Λετωνία οι ψηφοφόροι μου έχουν ένα πρόβλημα με τις άμεσες πληρωμές. Όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 οδηγηθήκαμε σε κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας. Εφτάσαμε να έχουμε το 14% το 40% συγγνώμη, το, το όσο είχαμε στην ε, προηγούμενη περίοδο, στη σοβιετική δηλαδή περίοδο. Λαμβάνουμε το 35% των του μέσου όρου των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα ΚΑΠ 20 πριν από λίγα χρόνια και οι γεωργοί μας θεώρησαν ότι θα καταργηθούν τα ιστορικά κριτήρια τώρα και θα αντικατασταθούν από άλλα καλύτερα. Για δύο χρόνια εμείς αγωνιστήκαμε και στην Επιτροπή αλλά και σε, άλλες, και σε άλλα βήματα. Στο επίπεδο των συζητήσεων τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά όταν ερχόμαστε στις συγκεκριμένες πληρωμές βλέπουμε τα πράγματα παραμένουν ίδια και απαράλλαχτα. Και οι ψηφοφόροι μου δεν το καταλαβαίνουν. Το 2020 θα φτάσουμε να έχουμε χώρες που θα λαμβάνουν μονάχα μόνο το μισό από το μέσο όρο της Ένωσης και άλλες χώρες θα έχουν το τριπλάσιο του μέσο όρου. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Οι ψηφοφόροι μου ζητούν να κάνω κάτι. Δεν δέχονται ότι μπορεί τα πράγματα να είναι σωστά. Υπάρχουν κατά τη γνώμη τους λόμπι τα οποία εδώ δίνουν χρήματα και με τον τρόπο αυτό εξαγοράζουν καλύτερες συνθήκες για αυτά τα ίδια. Τίθεται και το ερώτημα τι κάνουμε εδώ ως βουλευτές δεν επιτρέπει να υπάρχουν λόμπι. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, υπάρχουν ομάδε εργασία. Όργανα τα οποία επηρεάζουν τι εργασίε μα. Αυτό όμως θα πρέπει να το πιστέψουν οι ψηφοφόροι μας ότι είναι σωστό και αληθές. Δεν μπορούμε να προφασιζόμαστε ότι δεν έχουμε χρήματα. Εάν παίρνουμε από τον έναν και δίνουμε στον άλλο, αυτό δεν είναι δίκαιη λύση. Πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο των κοντιλίων που πηγαίνει, ποιος έχει συνεισφέρει πόσα και θυμούμε ακόμα τι το τότε. Ναι, μεν υπάρχουν ιδιωτηρότητες, αλλά δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από το 80% του μέσου όρου και πάνω από το 120% του μέσου όρου. Αυτά ίσως να μην αρέσουν σε ορισμένου, αλλά είναι σημαντικά για τις βαλτικές χώρες και για την Πολωνία. Αλλιώς θα προκληθεί η εντύπωση ότι την εξουσία εδώ την μοιράζονται μονάχα οι μεγάλες ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο. Πόσο καιρό θα τα συζητάμε ακόμη αυτά. Εγώ σας είπα εδώ και δύο χρόνια παλεύω και δεν έχει αλλάξει τίποτε. Αυτά πρέπει ωστόσο να λυθούν υπόψη. Μικρές χώρες και μικροί αγρότες, μικρές εκμεταλλεύσεις και αυτοί πρέπει να έχουν το δίκιο τους. Στην τελευταία ολομέλεια είπαμε ότι θα είμαστε ισχυροί μόνο όταν θα σκεπτόμαστε και θα φροντίζουμε όλους. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιξ. Ο σέρζο Σιλβέστρης και μετά ο Αντιπρόεδρο Μποφέ. Ε, ευχαριστώ. Σε συγχαίρω. Σας συγχαίρω για την εκλογή σας και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση σε δείπνο απόψε. Μας καλέσατε να το γιορτάσουμε με τυπικά ιταλικά προϊόντα. Ε, πρόκειται για πλάκα, για αστείο πρόκειται, λέει ο πρόεδρος Θημιδία στην Επιτροπή. ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σιλβέστρη. Αναφέρθηκε κάτι το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο σε όλους ότι ένα σωρό κριτικές ακούστηκαν αλλά ελάχιστε προτάσεις μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι από τις κριτικές που ακούστηκαν μέχρι σήμερα θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να ασκήσουμε σε βάθος το ρόλο που μας προσδίδει η συνθήκη της Λισαβόνας. Για τις άμεσες πληρωμές ο συνάδελφος Κάπουλα Σάντος είπε ότι για όποιον χάνει είναι δύσκολο να δεχθεί αυτούς τους όρους. Όποιος χάνει αρχίζει και διαμαρτύρεται. Σύμφωνοι, αλλά μιλάμε εδώ για απώλεια ε, όχι μόνο μίας καλλιέργειας αλλά ένας, ενός μεγάλου κομματιού της επικράτειας. Με τους λογαριασμούς που έχουμε διαπιστώνουμε ότι θα φτάσουμε σε άμεση πληρωμή που δεν θα ξεπερνάει τα 325 ευρώ ανά εκτάριο. Βασικές πληρωμές, πληρωμές greening όπως και επιπλέον οι συνδυασμένες πληρωμές ε, νέων κλπ. Ε, νέων ε, γεωργών κλπ. Κοιτάστε, εμένα η περιοχή μου που είναι κυρίως λιόδεντρα και ντοματιές έχουμε μέσες ε, τιμές της τάξης των χιλίων ευρώ. Άμα περάσουμε στα 325 είναι καταστροφή. Δηλαδή όταν έχουμε εμεί μία δραστηριότητα ε, αιωνόβια σε μία επικράτεια δεν μπορούμε να την αποδυναμώσουμε, δεν θα έχει πια καμία δύναμη για να συνεχίσει και δεν είναι κάτι το οποίο συνδέεται με ένα ή δυο ε, γεωργικές επιχειρήσεις. Μιλάμε εδώ για ολόκληρη η ανθρώπινη παρουσία στην επικράτεια. Διότι εμείς με αυτές τις επιδοτήσεις έχουμε ένα ολόκληρο δίκτυο στην, στην περιοχή, δηλαδή δεν έχουμε μόνο λιόδεντρα. Έχουμε ελαιοτριβία, έχουμε εργοστάσια μεταπικοσερβοποίησης της ντομάτας. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα σκεφτούμε όχι υπό την έννοια ότι παραπονιέται κάποιος γιατί χάνει, αλλά γιατί ολόκληρα τμήματα της επικράτειας δεν μπορούν πια να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και όπου η Ένωση μέχρι χθες, μέχρι σήμερα συνέχιζε να επενδύει. Ζητούμε αντικειμενικά επιπλέον μέτρα για τον υπολογισμό της άμεσης βοήθειας, ε, για το ακαθάριστο πολιτε, ε, πολιτεοπροϊόν, δεν θα πρέπει εμείς μέσα από την κατάργηση των άμεσων πληρωμών να κρεμίσουμε όλο το δίκτυο το οποίο έχουμε διαμορφώσει ως σήμερα για τους ενεργούς τώρα γεωργούς και τον ορισμό τους. Ένα άλλο από τα έξι σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο εισηγητής είναι αδιανόητο να μην δίνουμε πόρους μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Φυσικά και πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς που ζουν από τη Γεωργία. Αλλά ας λάβουμε και άλλα κριτήρια υπόψη μας στον ορισμό ενός ενεργού Γεωργού. Πιο ευθύγραμμα, πιο λογικά από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Ας δούμε ποια είναι τα, ποιος είναι ο τζίρος των επιχειρήσεων. Να δούμε τι διοχετεύουν στην αγορά αυτές οι επιχειρήσεις. Να θεωρήσουμε ένεργο τον Γιωργό ο οποίος παράγει και δυσδιεί στην αγορά. Αυτός είναι ο στόχος της ΚΑΠΑ, είναι να εγκιάται την τροφιμική ασφάλεια. Ας δούμε επίσης και την δυνατότητα για την εκτιματική αναδιάρθρωση εμείς στην Ιταλία μοιράζουμε τις άμεσες βοήθειες ανάλογα με τα εκτάρια και έχουμε κόσμο ο οποίος παίρνει χίλια, λιγότερα από χίλια ευρώ ή ακόμη έχουμε και επιδοτήσεις κάτω των 500 ευρώ. Δεν μπορούμε εμείς να υποστηρίζουμε μόνο αυτούς οι οποίοι κάνουν οικογενειακή γεωργία, πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς που κάνουν έρευνα, που παράγουν προϊόντα που πάνε στην αγορά και συνδράμουν ε, στον στόχο της αυτάρκειας. Εμένα στην περιοχή μου συνεχίζουμε να δίνουμε το να το πριν σε νέους γιοργούς, 20.000 ευρώ κτλ όπου αυτοί οι νέοι παίρνουν τις ε, ε, εγκαταλελειμμένα χωράφια των γονιών τους. Το θέμα λοιπόν της ε, κτηματολογικής αναδιάρθρωσης πρέπει να αποτελεί στόχο για να μπορέσει να είναι η γεωργία μας στη σύγχρονη αγορά, να επενδύει και να καινοτομεί. Για το greening, εμένα μου φαίνεται ότι αντί να διευκολύνουμε την ζωή των καλλιεργητών, τους την μπερδεύουμε με νέους ορισμούς, με νέες γραφειοκρατίες, με νέες αρμοδιότητες που σήμερα οι γεωργικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να, το αντέξουν. Η υπερβολή της ε, γραφειοκρατίας δεν μπορεί να, να, να έρθει και με τη νέα ΠΑΚ. Ε, κοιτάστε, τι γίνεται. Ένας ελαιώνας ε, πόσο διοξίδιο του άνθρακος απορροφά σε σχέση με ένα μποσκότοπο και δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί η συμβολή του ελαιώνα στην μείωση του διοξιδίου του άνθρακος και άμα κάνει και βιολογική γεωργία δεν θα πρέπει να... Δεν θα πρέπει να αποζημιώνεται άμα ε, υπάρχει μια κήτη ποταμού στην εκμετάλλευση, στη γεωργική εκμετάλλευση, δεν θα πρέπει και αυτό να ενισχύεται, να αποσημειώνεται. Υπάρχουν απλοί στόχοι λοιπόν. Ευχαριστώ Σέρτζο. Ο Αντιπρόεδρος Μποβέ και μετά κυρία Ρανσκασία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που ανανεώσαμε το Προεδρείο μα, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι να είμαστε πάλι εδώ. Τώρα επειδή όμω είμαστε στην αρχή τη περίοδου αυτής και έχουμε δυόμιση χρόνια να εργαστούμε μπροστά μα για την ΚΑΠ, πρέπει να πω ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα όταν εργαζόμαστε για την ΚΑΠ να είμαστε ανεξάρτητοι έναντι το λόμπι και όλων εκείνων που θέλουν να υποστηρίξουν κάψουν τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να την υποβάλψουν σε μεγάλα συμφέροντα στην ε, βιομηχανική βιομηχανία γεωργικών φαρμάκων ή στην ε, ε, μηχανική γεωργία. Για την έκθεση Καπούλα Σάντος θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Πρέπει να μπούμε εμεί στη λεπτομέρεια των κειμένων και πρέπει να τα αναλύσουμε διαπιστώνουμε στα σχόλια να υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε στο κείμενο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην λέμε ότι θέλουμε να σταθώ σε μερικά. Δεν θέλω να συζητήσω για τη φιλοσοφία του πράγματος, τη φιλοσοφία ήδη τη συζητήσαμε. Για τη χρηματοδότηση των κρατών μελών και την πανεξισορρόπηση των κρατών μελών. Εμείς έχουμε πρόβλημα όταν βλέπουμε τις προτινόμενες τιμές για την κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Λέμε λοιπόν ότι αν οι χώρες αυτές έχουν μία διαφορά με 80% ε, διαφορά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τότε ε, ε, ίσως και Αλλά τι γίνεται όμως όταν μια χώρα έχει 75% για να μπορέσει να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους, θα μας χρειαστούμε χρόνια και χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να φτάσουμε στο 2048 για να έχουμε την ισορροπία. Δεν λειτουργεί λοιπόν. Έχουμε πρόβλημα. Το επισημένο. Αυτό για την ισορροπία μεταξύ των χωρών. Δεύτερο πρόβλημα. Με τους ενεργούς γεωργούς συμφωνούμε με τη φιλοσοφία. Οι ενεργοί γεωργοί πρέπει να είναι αυτοί που αποζημιώνονται. Αλλά να δούμε τα νούμερα τα οποία προτάθηκαν σχετικά με το κατά πόσο δηλαδή το ποσό των άμεσης, βοήθειας ε, είναι 5% κάτω από τα έσοδα. Αν έχουμε τώρα τη βασίλισσα της Αγγλίας, όχι για να της επιτεθώ, καλή γυναίκα είναι, η οποία παίρνει 300.000 ευρώ βοήθεια. Άμα ξεπερνάει λοιπόν τα 6 εκατομμύρια το χρόνο, παίρνει τα 300.000 χιλιάρικα. Αν όμως κερδίζει 5.999 ευρώ, τότε τη βοήθεια την παίρνει. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα εξετάσουμε πιο σωστά. Θεωρητικά και πρέπει να το διευκρινίσουμε, άμα δούμε καλά το κείμενο, οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να παίρνουν βοήθεια. Πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είδαμε για τις ε, ζάχαροβιομηχανίες ή για τις μεταφορικές εταιρείες δημητριακών ή ζωών που ενισχύθηκαν ε, και έχω κατά νου την Κάργιλ. Πρέπει να τα προσέξουμε. Για τους γεωργούς λοιπόν δεν επανέρχομαι, για την ε, πτωτικότητα δεν έχω να πω τίποτα. Να σταθώ και σε κάτι άλλο πρέπει να μιλήσουμε για τις αγροπεριβαλλοντολογικές ενισχύσεις. Εγώ πιστεύω ε, ότι επισημάνθηκαν προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι τα προβλήματα δεν αποτελούν φάντασμα. Όταν εμείς λέμε ότι το 7% των εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να αποτελούν ε, ε, επιφάνειες ε, οικολογικού ενδιαφέροντος. Δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να είναι περιοχές οι οποίες έχουν μείνει σε αγρανάπαυση. Εγώ νομίζω ότι σε μια γεωργική εκμετάλλευση όπως κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ των, ε, των γεών οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες και εκείνες οι οποίες ε, δεν καλλιεργούνται. Είναι ένα κριτήριο που είναι περίεργο. Για να έχουμε αυτό το 5% τι σημαίνει. Θα πάρουμε εμείς ε, τις, ε, τους, ε, το, τους τείχους από φυτά, θα πάρουμε τους, τα κτίσματα, πώς θα το δούμε αυτό. Η αρχή είναι καλή, αλλά αυτό το οποίο θεωρώ επικίνδυνο είναι ότι δίνουμε μέχρι το 2014 την δυνατότητα αλλαγή προορισμού αυτών των γεών. Δηλαδή η διάταξη του 2014 θα ορίσει τα κριτήρια. Μέχρι το 2014 μπορούμε να έχουμε τροποποίηση στις χρήσεις των γεών. Αυτό μου φαίνεται επικίνδυνο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία επιτάχυνση αύξηση των βοσκοτόπων. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε ένα μέσο όρο πολλών ετών, αλλά όχι μία οριστική χρονιά στα δύο ή τρία χρόνια, γιατί αυτό θα μπορούσε να έχει το ανάποδο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε, για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και τελειώνω. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. 70% ε, μεγαλύτερη επιφάνεια, μικρότερη 5%. Δεν μιλάμε για τις φυτικές πρωτεΐνες και για την κύκλωση των, την κυκλωτική καλλιέργεια. Η ΚΑΠ δεν είναι μόνο γραφειοκρατία για να δίνει λεφτά, στοχεύει και στον προσανατολισμό της γεωργίας προς μια κατεύθυνση. Το ψηφίσαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, το θέμα της κυκλωτικότητας των καλλιεργιών. Και η αυτονομία σε φυτικές πρωτεΐνες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί. 70% σε μία ενιαία καλλιέργεια, έχουμε μόνο καλλιέργεια και δεν έχουμε αγρονομία. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν διευκρινήσεις σχετικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέρεντς Γκαρσία. Πολλοί από εμά δεν συμφωνούμε με το θέμα, αλλά γιατί φαίνεται να εξαφανίζεται ένα ιστορικό κριτήριο στην ΚΑΠ. Θα έπρεπε λοιπόν να λάβουμε η υπόψη μας ότι μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα τραυματικές καταστάσεις και θα έπρεπε κύριε Κάπουλας και ορισμένες ειδικέ μεταβατικές διατάξεις για αυτούς, διότι έτσι θα πλήξουμε ορισμένους τομείς όπως τον τομέα των ζωοτροφών που θα ζημιωθούν, όπως επίσης τον τομέα ελαιολάδου ή του ρυζιού, της οριζοκαλλιέργειας που υπέστησαν και πρόσφατα ζημιές. Για αν θα αποφύγουμε εμείς ε, την ολική περικοπή των επιδοτήσεων σε αυτές, για αυτές τις καλλιεργίες, τότε θα έπρεπε να αποφασίσουμε κάποια άλλα ειδικά μέτρα. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα, χεριστά, τα χωριστά μοντέλα παραγωγής στην πρόταση. Ας πούμε, το θέμα της κτηνοτροφίας χωρίς ε, ε, ε, συγκεκριμένη χωροταξική βάση επίσης ε, δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα οι συνδυασμένες ε, πληρωμές σε αυτόν τον τομέα συνδέονται και με άλλα είδη κτηνοτροφίας και δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε αυτή την κτηνοτροφία χωρίς βοήθειες. Θα ζημιώσουμε τομείς που θα έπρεπε να, έπρεπε να υποστηριχθούν. Το τρίτο σημείο, επιλέξιμα εκτάρια. Εμένα μου έρχεται πανικός ε, όταν σκέφτομαι ότι αυτό θα μπορούσε να είναι καπές για όλους. Και θα αυξηθούν ε, τεράστια τα εκτάρια που θα ζητηθούν από τα κράτη-μέλη. Επειδή είμαστε περιορισμένοι στον προϋπολογισμό και επειδή δεν έχουμε ε, δυνατότητες. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σε... σεβάσμοι έναντι των παραγωγών και των χρηματοδοτήσεων που τους δίνουμε. Πρέπει επίσης να υπάρξει ένας δεσμός μεταξύ παραγωγικής βοήθειας και της χορήγησης των ενισχύσεων. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πώς θα αλλάξουν όλα αυτά. Εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός Ε, της υποχρεωτικότητας. Τώρα για το greening, εγώ πιστεύω ως, ε, ως Ισπανίδα, ε, πιστεύω ότι αυτή η λογική του greening λαμβάνει υπόψη της εκτάσεις στην κεντρική ή στη Βόρεια Ευρώπη. Μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη με τίποτα οι τοπικές πραγματικότητες όπως για παράδειγμα η πραγματικότητα στο Νότο. Θα ήθελα ε, να πω άλλα δύο πράγματα και τελειώνω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε την διπλή χρηματοδότηση, διότι στο παρελθόν είχαμε για το ίδιο σχέδιο δύο παράλληλες ε, μορφές χρηματοδότησης και μείναμε ε, χωρίς τίποτα στο χέρι στο τέλος θα πρέπει να έχουμε στον πρώτο πυλώνα τις άμεσες βοήθειες που έχουν να κάνουν με τα ε, φυσικά προβλήματα και το δεύτερο, το δεύτερο πυλώνα να τον θέσουμε με την παραγωγικότητα. Τώρα, για την κατάργηση των ποσοστώσεων του, του, της ζάχαρης. Το 2004 εγκρίναμε και εφαρμόσαμε από το 2007 μία δραματική μεταρρύθμιση όπου χάθηκαν πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζαχαρότευλων στην Ιβυρική Χερσόνησο. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδού και οι ποσοστώσεις πρέπει να κρατηθούν μέχρι το 2020. Πρέπει να συγχαρώ επίσης τον Επίτροπο, ο οποίος ανακοίνωσε ε, την, ε, την συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας η οποία συζητάει για τα δικαίωμα φύτευσης αμπελώνων. ο κύριος Ταραμπέλα. Πολλά πράγματα υπόθηκαν ήδη κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πλέον απόδειξη ότι πέρα από τις πολιτικές μας ζυμώσεις υπάρχουν πράγματα τα οποία τελικά, με τα οποία τελικά συμφωνούμε. Και όπως το κάναμε με την έκθεση του George Lyon και μετά με την έκθεση Des, πρέπει να προσπαθήσουμε να βγει από το Κοινοβούλιο ένα σαφές μήνυμα. Διότι είχαμε μία μικρή εμπειρία μεταξύ του τριολόγου και του κυρίου κύριο Όλσον ο οποίος θέλησε να μας μαζέψει όλους, ε, τον κύριο Ράιμερ, τον κύριο Φοντάνα και δεν ξέρω ποιον άλλον ε, και διατυπώσαμε προτάσεις οι οποίες έτειναν προς έναν κοινό στόχο. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι ο αντίπαλός μας είναι το Συμβούλιο. Και όταν το λέω αυτό, γιατί, γιατί το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα διαιρεμένο, διότι ε, ταμπουρώνεται πίσω από τις εθνικές θέσεις πολύ περισσότερο από μας. Και προσοχή όταν θα υπάρξει τρίλογος... Το Συμβούλιο μπορεί να έρθει εδώ χωρίς εντολή, διότι υπάρχει η ε, ε, μειοψηφία τροχοπέδησης η οποία το εμποδίζει να, να προβάλλει θέσεις. Και σε επίπεδο κοινοβουλίου μας έχουν έρθει μηνύματα σχετικά και αν συνεχίσουμε προς την ίδια γραμμή που συνεχίζουμε θα ήταν πολύ θετικό. Εγώ δεν θα μιλήσω για όλα. Αλλά δεν είμαι υπέρ της εξέλιξης ε, μιας ενιαίας πληρωμής δηλαδή στο μέλλον ανεκτάριο. Αυτό σημαίνει ότι αγνοούμε με αυτό, το, αυτό το οποίο κάναμε μέχρι τώρα. Διότι εμείς ανερούμε την, ε, τους στόχους της Γεωργίας. Μια τέτοια πολιτική σημαίνει ότι εντάξει αγνοούμε τους στόχους και σας δίνουμε ούτως ή άλλως παράδες. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε το 2020 λέγοντας πάρτε τόσα γιατί είχατε το 2003 άλλα θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια για τον Γιωργό, άντρα γυναίκα, ε, για την επίτευξη στόχων. Διότι τελικά τι γίνεται όταν έχουμε εμείς ενιαίες πληρωμές σημαίνει ότι χρηματοδοτούμε τους γεωκτήμονες, και όχι, δηλαδή την αξία της γης και όχι τη δουλειά του αγρότη της αγρότησας. Εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε ιδιαίτερες πιέσεις στην παραγωγή και αυτό λόγω της παραγωγής γεωκαυσίμων. Τώρα, γεωργική δραστηριότητα παντού, σύμφωνη. Θα πρέπει όμως να είναι συνδυασμένη. Αυτό το 5% είναι ανεπαρκές για ορισμένες περιφέρειες. Άμα πάρω εγώ τώρα την Βαλονία εδώ στο Βέλγιο, είμαστε στο 20%. Προσοχή λοιπόν, με τέτοιου είδους μηχανιστικά νούμερα ε, στρεβλώνουμε την πραγματικότητα σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης όπου θα ήταν καλό να διατηρήσουμε μία γεωργική δραστηριότητα συν τις μεταποιητικές ε, δράσεις σε όλη την περιοχή. Τρίτο, πρέπει να συμβάλλουμε να έχουμε μία γεωργική δραστηριότητα η οποία ε, ευεργετεί όλη την κοινωνία. Εντάξει το greening, αλλά έχουμε και τα public boots ε, σε δεύτερο ή στον τρίτο πυλώνα, θα δούμε. Το 7% προσοχή, μην είστε τόσο μαθηματικοί. Λοιπόν, η Αυστρία είναι ένα μοντέλο. Το 90% των γεωργών έχει εγκρίνει τα αγροτροφημικά μέτρα. Είναι πρωτοπορία η Αυστρία στις βιολογικές καλλιέργειες. Δεν ξέρω, δεν θα έπρεπε να πάμε εμείς αγρόκτημα προς αγρόκτημα, αλλά θα έπρεπε ίσως να το ορίσουμε χώρα προς χώρα. Το να πάμε, πηγαίνουμε εμείς αγρόκτημα προς αγρόκτημα μου φαίνεται ιδιαίτερα μηχανιστικό. Και ξέρετε, εγώ είμαι κατά της της γραφειοκρατίας, αλλά το διοικητικό σκέλος είναι πάντοτε χρήσιμο. Τώρα, γεωργή, ενεργή γεωργή, πρέπει οπωσδήποτε να το επανοπροσδιορίσουμε. Υπάρχουν ακόμη πολύ σύμφωνα με τον ορισμό της Κομισιόν ε, όπου υπάρχει ένας σωρός κόσμος ο οποίος δεν ασκεί γεωργική δραστηριότητα αλλά θεωρείται ενεργός γεωργός. Λοιπόν, το θέμα της σταδιακής πτώσης, ε, όλα αυτά τα είχε θέσει το Κοινοβούλιο, ας το ακολουθήσουμε στο μέλλον, αυτό μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και άμα οδηγηθούμε και στην αποκατάσταση υπηρεσιών, ε, ισορροπιών, συγγνώμη, μεταξύ μεταξύ των διαφόρων ε, περιοχών της Ευρώπης. Τώρα η Λετωνία ίσως να διαπραγματευτεί και άσχημα και παίρνει 60 ευρώ ανά εκτάριο όταν η Μάλτα παίρνει 60 600 ε, ε, συγγνώμη η Ολλανδία παίρνει 500 πρέπει να δούμε εμεί όμως ποιοι είναι οι στόχοι και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία όμως θα πρέπει να επαναξισορροπούν τις ενισχύσεις υπάρχει όμως ένα βασικό σημείο είναι τι κάνουμε για τη ρύθμιση των αγορών. Η πρόταση νομίζω ότι δεν είναι αρκετά ισχυρή, δεν εμπλέκει επαρκώ στον δημόσιο τομέα. Ο Μισελ Νταντέν θα μας τα πει αυτό με όταν θα μιλήσει σχετικά με τις ΚΟΕΣ, τη κοινή οργάνωση αγοράς. Χαμογελάει ο Ζωζεμποδέ, δεν ξέρω γιατί. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα μοντέλο όπου ο καθένας ε, ε, εμπλέκεται αλλά υπό το καπέλο των αρχών. Και αν εσείς αυτό το λέτε γραφειοκρατία, εγώ είμαι υπέρ της γραφειοκρατίας τότε. Θα πρέπει να έχουμε δηλαδή χωροφύλακες που θα πρέπει να ορίζουν ποια είναι η δίκαιη τιμή και ποια δεν είναι διότι εμείς μιλάμε για εισόδημα γεωργών ανδρών και γυναικών, σίγουρα μέσα από τις ενισχύσεις, αλλά κυρίως μέσα από τη σωστή αμοιβή για όλους τους αγρότες και αγρότησες σε κάθε από τις μια παραγωγές. Υπάρχει λοιπόν πολύ νερό στα βλάκια. αναγνωρίζω στην Κομισιόν ότι θέλησε να ερμηνεύσει προτάσεις και ανησυχίες του Κοινοβουλίου δεν μπορούμε εμείς να τους το προσάψουμε. Αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ, να εξετάσουμε καλύτερα ορισμένα κεφάλαια για να συνεχίσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να στέλνουμε σαφή μηνύματα και να μην έχουμε δηλαδή μία άγευστη μεταρρύθμιση, αλλά μία μεταρρύθμιση που θα προστατεύει όλων των τύπων της γεωργίας συνδυάζοντας με καλύτερη διαχείριση του νερού, με τη διαχείριση του εδάφους, προστατεύοντας δηλαδή το περιβάλλον. Το Συμβούλιο όμως δεν έχει αυτή τη λογική. Πρόκειται για έναν συνδυασμό εθνικών συμφερόντων. Θέλουμε εμείς η ΚΑΠ να αποτελεί πραγματική μεταρρύθμιση που θα προσεγγίζει τους στόχους που έχει θέσει ήδη αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Μάρκ. Ντότς και μετά Σκότα. Ευχαριστώ και από εμένα συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Πρώτα, ευχαριστώ και τον εισηγητή για τα σχόλιά του στην αρχή της συζητήσεως. Η συζήτηση μέχρι τώρα δείχνει πόσο ευαίσθητη θα είναι η διαδικασία. Η συζήτηση γυρίως για τις άμεσες πληρωμές που θίγει ορισμένες από τις ευαισθησίες που σημειώνονται σε όλες τις συζητήσεις μας τα τελευταία χρόνια. Όταν ψηφίσαμε την έκθεση ΛΑΙΟΝ ψηφίσαμε βέβαια υπέρ μιας δίκαιης κατανομής, που αυτή δεν σημαίνει βέβαια ίση κατανομή, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και κόστος παραγωγής, αξία γης κλπ. Βεβαίως θα αναφέρω πράγματα που ενδιαφέρουν την ε, εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια, Βόρεια Ιρλανδία. Έχω συζητήσει και με Σκότους συναδέλφους μου. Ορισμένοι από που έχουν, ε, ορισμένα τα προβλήματα που έχουν σημειώνονται και στη δική μου εκλογική περιφέρεια, τη Βόρεια Ιρλανδία. Εμεί έχουμε ένα υβριδικό σύστημα πληρωμών με ιστορικά στοιχεία για μεμονωμένες δηλαδή αγροτικές εκμεταλλεύσεις, single farm payments, οι γεωργοί μας όταν μιλώ μαζί τους εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την ταχεία κίνηση που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ένα σύστημα κατά flat rate. Εάν για παράδειγμα πάμε στο 40% το πρώτο έτος, το έτος 1, αυτό μοιραία θα οδηγήσει ορισμένες εκμεταλλεύσεις εκτός αγοράς, θα τις διώξει από τη δουλειά πολλές από τις εκμεταλλεύσεις αυτές είναι εντατικής, ε, εντατικών συστημάτων και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Εγώ ζητώ μάλιστα παράταση της προθεσμίας του 2019, διότι όπως είπατε και εσείς στις αρχικές σας παρατηρήσεις, δεν επιτρέπεται να ανατρέψουμε τις εθνικές ισορροπίες σε τρόπο που να οδηγήσουμε σε καταστροφή τους ντόπιου γεωργούς. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει εδώ λόγος μεγάλης ανησυχίας για τους ε, αγρότες της Βόρειας Ιρλανδίας. Στη Βόρεια Ιρλανδία το σύστημά μας είναι επίσης περίπλοκο, το κόνικερ, το οποίο είναι ένα είδος ε, μίσθωσης της γης. Ένα τρίτο της παραγωγής μας είναι ωστόσο από μισθωμένη γη για σύντομα χρονικά διαστήματα και γι' αυτό μας, οδηγεί, ε, γι αυτό σε αυτό το σύστημα το Single Farm Lane ε, το Single Farm γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει θα πηγαίνουν τα χρήματα στην εκμετάλλευση όπως και φορέας της ή σε αυτόν που έχει την άδεια λειτουργίας. Η Κομισιόν θα πρέπει να διευκρινίσει ακριβώς ποιος είναι ο δικαιούχος για την συγκεκριμένη πληρωμή. Είχαμε και ένα πρόβλημα στην Ιρλανδία Πολλά από τα σενάρια της πρότασης επιφέρουν σημαντικές δυσκολίες. Και έρχομαι στην έννοια του ενεργού αγρότη. Πώς θα μετρώνται τα ε, σχετικά κριτήρια μέσα στο χρονικό πλαίσιο. Υπάρχουν περίπλοκα ερωτήματα λοιπόν και για τη Βόρεια Ελλανδία συνδέονται και με τη μίσθωση της γης. Για το greening πάλι αυτό προκαλεί σημαντικά προβλήματα σε εμά στη Βόρεια Ελλανδία. Το 90% της γης είναι βοσκοτόπια. Θα έχουμε λοιπόν ορισμένα πλεονεκτήματα από ορισμένα, βεριατήματα μάλλον από τα μέτρα για το πρασίνισμα, αλλά υπάρχουν και ορισμένες αρρώσιμες γέες, οι οποίες με την διαφοροποίηση της εναλλαγής των καλλιεργειών θα οδηγηθούν σε μειονέκτημα. Και δεν θα μπορούν πλέον να ε, καλλιεργούν αρρώσιμες γέες. Επίσης, βγάζοντας το να βγάλει κανείς το 7% για το set aside πρόγραμμα των γεών, πάλι αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή μου. Αυτό σημαίνει ότι υπονομεύεται το βασικό στόχος της ΚΑΠ, δηλαδή η παραγωγή τροφίμων, καθώς επίσης μειώνει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Οι προτάσεις είναι περίπλοκες. ιδιαίτερα για το πρασίνισμα όπου σημειώνονται, θα υπάρξουν και προβλήματα από τη γραφειοκρατία και για τα βοσκοτόπια εγώ πήγα στα Uplands στην περιοχή κοντά στην βόρεια ακτή μας σε ένα όμορφο μέρος της ε, εκλογικής μου περιφέρειας και συνομίλησα με τους αγρότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα σχετικά με τα μόνιμα βοσκοτόπια και τι επιτρέπεται να κάνει κανείς μέσα σε αυτά τα και για παράδειγμα εάν εκεί όπου φύονται οι πόες είναι ε, δυνατόν να γίνεται να θεωρηθεί ως βοσκοτόπι ή πρέπει να είναι ή μπορεί να είναι και αρρώσιμη γέα. Εάν λάβουμε υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, αυτό είναι απαραίτητο γιατί τότε θα επιτρέψουμε στους αγρότες να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ, Ντότς. Σκότα και μετά Άλμπερτ Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτα, πολλές ευχές για όλες και όλους, για την καλή χρονιά. Ακούγονται πολλές ερωτήσεις ε, στην, ε, στην Ήπεθρο και θέλω να τις αναφέρω εδώ. Οι Γεωργοί θεωρούν ότι κάπως ιδιάζουσα η διάταξη του άρθρου 21 όπου θεωρείται το 2011 ως έτος αναφοράς για την χορήγηση της βασικής πληρωμής και αποκλείονται οι κατηγορίες εκείνες των γεωργών που του 2012 ή το 2013 είχαν το δικαίωμα των ενιαίων επιδοτήσεων. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να αποφύγει την κερδοσκοπία ο νομοθέτης, σύμφωνοι. Από το 2013 όμως αυτή η διάταξη θα έπρεπε να τροποποιηθεί ούτως ώστε να συμπεριληφθούν εκείνες οι κατηγορίες που αποκλείονται. Και αναφερόμαστε εδώ στους ενεργούς γιοργούς. Να καταλάβουμε αν ο ενεργός γιοργός είναι το βασικό, ο βασικός δικαιούχος αυτών των άμεσων πληρωμών. Ευχαριστώ Τζανκάρλο. Ο κύριος Ντες και μετά Ανιού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας συγχαίρω και για την επανεκλογή σας. Συγχαρητήρια και στους ε, αναπληρωτές. Ε, ε, προσβλέπουμε στην συνέχιση της καλής συνεργασίας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καπλασάντος ε, για τις πρώτες του παρατηρήσεις μια επίκριση δεν ήταν ε, αρκετά αναλυτικές ε, οι παρατηρήσεις σας και εγώ όταν ξεκίνησα με κατηγόρησαν ότι δεν ήμουν αρκετά αναλυτικός. Ε, απ' την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπερβάλλει κανείς και στις ε, λεπτομέρειες. Έχουμε χρόνο για να πούμε στις λεπτομέρειες. Ε, είμαι πεπισμένος ε, ότι θα ακούσουμε ε, από τις πολιτικές ομάδες και από τους συναδέρφους αναλυτικές προτάσεις, οι οποίες φυσικά θα πηγαίνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Θα πρέπει από αυτές να επιλέξουμε τι είναι καλύτερο για τη γεωργία στην Ευρώπη. Και δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε τι είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο τι, ε, και, τι, και τι μπορούμε να πληρώσουμε. Στην... Στο Βερολίνο βρεθήκαμε ε, στις εκδηλώσεις για την Πράσινη Εβδομάδα. Ε, τελικά δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε ε, γεωργική πολιτική όπου οι γεωργοί να λαμβάνουν 20% λιγότερα χρήματα αλλά να πρέπει να έχουν 20% περισσότερη γραφειοκρατία. Ε, με ενοχλεί κάπω η πρόταση της Κομισιόν, διότι εάν παραμείνει ως έχει θα οδηγήσει σίγουρα σε περισσότερη γραφειοκρατία. Ως ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις απλοποίησης ε, χωρίς να ξεχάσουμε τον στόχο της γεωργική πολιτικής και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. με την έκθεσή μου μπορούμε να παρακαλέσουμε την ε, Κομισιόν ε, να μην ε, επιβάλλει περαιτέρω ελέγχου. αν υπερσφυριστεί με 90% μια έκθεση δεν είναι πια δική μου, είναι του Κοινοβουλίου. θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι τέτοιο από την Κομισιόν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές στα διάφορα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με τον το συνάδελφο Ρούμπιξ ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε το εξής. κατόπιν ε, πρόσκληση σε συναδέρφου, ε, Αγγλίδα συναδέρφου, είδα την κατάσταση επιτόπου. Δεν θα επιτρέπεται μετά το 2014 να έχουμε διαφορά ανάμεσα στο 52% και το 100%. Θα πρέπει να έχει υπάρξει κάποια ε, εξίσωση. Δεν... Ε, Θα πρέπει να ε, φτάσουμε σε μεγαλύτερες εξομοιώσεις ε, για λόγους ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Και θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί. Είτε μιλάμε για την Πορτογαλία, είτε μιλάμε για την Βουλγαρία, υπάρχουν σχετικά ε, πολλά χρήματα στον δεύτερο πυλώνα. Για διάφορους λόγους όμως δεν μπορεί πάντα να γίνει συγχρηματοδότηση και θα πρέπει να εξετάσουμε την ανακατανομή από τον δεύτερο στον πρώτο πυλώνα, κάτι που ξεπερνάει ε, τα πλαίσια της πρότασης ε, της Κομισιόν. Ε, αν μεταφέρουμε πόρους από τον δεύτερο πυλώνα στον πρώτο, τότε θα έχουμε μια εξημείωση. Πέρσι, κατά την Πράσινη Εβδομάδα, η Υπουργό Γεωργία τη Γερμανία είπε ότι η Γερμανία είναι διατεθειμένη να επιδείξει περισσότερη αλληλεγγύη ε, και μάλιστα να ε, ε, παραιτηθεί από κάποιες άμεσες πληρωμές όχι τελείω βέβαια αλλά και η υπουργό συμφωνεί με κάποια μερική παρέτηση από τις άμεσε πληρωμές κάτι τέτοιο θα απλοποιούσε τα πράγματα. Στη συνεργασία λοιπόν με το Συμβούλιο θα πρέπει να βρούμε την ε, σωστή λύση. Όσον αφορά το θέμα του ενεργού γεωργού, ε, πέρσι ε, μίλησα με τον Φραντς Φίσλερ, ο οποίος μου είπε ότι επί 10 χρόνια προσπαθεί να βρει μια λογική λύση. Το πρόβλημα όμως ήταν πάντα ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Δεν ε, θα πρέπει μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μπορεί να μας πει ότι αγαπητό Κοινοβούλιο, αγαπητό Συμβούλιο, αποφασίσατε κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε ρυθμίσεις οι οποίες να στέκουν. Στην ε, δική μου ε, περιφέρεια λέμε ότι ο ενεργός γεωργός θα πρέπει να ε, λαμβάνει εκτόσεις σε πολλές εκμεταλλεύσεις έχουν 80% εκτάσεις αγρανάπαυσης. Αυτό δεν συνάδει με τον ορισμό του ενεργού γεωργού και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό κατά την όλη συζήτηση, αλλιώς ε, γελιοποιούμεθα με τις δηλώσεις μας περί ενεργών γεωργών ε, εάν το 80% ε, έχουν εκτάσεις αγρανάπαυσης. Όσον αφορά τη ρύθμιση με το 7% δεν ε, μπορούμε να έχουμε μία ρύθμιση για 40 εκατομμύρια γεωργούς ε, στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ε, προβλέψουμε δεσμευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες όμως να μπορούν και να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να υπάρξουν εκτόσεις σε περιφέρειες όπου δεν υπάρχει αρκετή δραστηριότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη απέναντι στον κάθε γεωργό της Ευρώπης και η πολιτική μου ομάδα θα ασχοληθεί εντατικά με το θέμα ε, στο μέλλον και θα έχουμε σίγουρα έντονες ε, συζητήσεις ε, ώστε μαζί με τα άλλα 26 κράτη-μέλη να ε, βρούμε μια κοινή γραμμή. Πάντως είμαι αισιόδοξο ότι αν υπάρχει καλή βούληξη θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια γεωργική πολιτική που να ωφελήσει και τον γεωργό και τον καταναλωτή. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση. Είμαι αρκετά αισιόδοξο. Ευχαριστώ. Uh, um, uh, And, um, at the moment, Hollis... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα καταρχήν να σας, ε, ε, να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας ε, εσείς και εγώ προερχόμαστε από ε, διαφορετικά άκρα του πολιτικού ράνιου τόξου. Εγώ είμαι από την δεξιά, εσείς από την αριστερά. Εγώ είμαι Βρετανός, εσείς όχι. Ε, φαντάζομαι ότι θα ε, εξοργίζεστε συχνά όταν με ακούτε να μιλώ, επειδή θα διαφωνείτε με όλα όσα λέω. Πάντα όμως ε, ακούτε με δίκιο τρόπο την ε, θέση μου και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι είσαστε ε, αμερόληπτος πρόεδρος πολύ σημαντικό και επίσης καταβάλλετε προσπάθειες να προφέρετε σωστά το όνομά μου το οποίο ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο όσον αφορά, ας πέρασουμε τώρα στο θέμα, όσον αφορά τις ε, πολλαπλές καλλιέργειες, ε, αυτό το θέμα είναι αποτυχία. Επί δυόμιση χρόνια βρίσκομαι ε, στην Επιτροπή τούτη και ακούω ανθρώπους ε, κυρίως από την αριστερά να λένε πόσο σημαντικό είναι η Επιτροπή μας ε, να στηρίξει τους ε, μικρούς ε, γεωργούς. Ε, αυτοί είναι οι άνθρωποι τους οποίους θα πρέπει να φροντίζει η κοινή γεωργική πολιτική. Όσον αφορά λοιπόν τις πολλαπλές καλλιέργειες, ας κοιτάξουμε την μικρή εκμετάλλευση κτηνοτροφίας και την μικρή εκμετάλλευση ερώσιμης γης. Αν έχουμε κτηνοτροφία, το 90% θα είναι βοσκότοποι. Μπορεί όμως να ένα μέρος ε, να ε, είναι αφοσιωμένο στην ε, καλλιέργεια κρυθαριού και Έτσι μπορούν να ταΐσουν τα ζώα και αυτό επίσης αποτελεί καλή βάση για να αποκατασταθεί ο σκότοπος, το χόρτο δηλαδή μετά από μερικά χρόνια. Αντί για κρυθάρι όμω θα πρέπει να έχουν τώρα τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τι άλλες καλλιέργειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Σκεφτήκαμε την, τη, βρώμη, ε, το έχω συζητήσει αυτό με μικρού γεωργούς. ναι, θα μπορούσε να πει κανεί ότι και η βρώμη είναι μια δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να αποθηκευθούν ε, αυτές οι ε, αυτές τις καλλιέργειες, ε, αλλά το κρυθάρι και η βρώμη θα πρέπει να αποθηκευτούν ξεχωριστά, το οποίο σημαίνει ε, επιπλέον κόστος. Επίσης μπορούν εύκολα να καλλιεργηθούν βιολογικά αυτές οι καλλιέργειες. Εάν όμως επιλέξουν άλλες καλλιέργειες, ε, είναι αρκετά ακριβώ ο σπόρος σε αντίθετη με τα προηγούμενα και επίση θα αντιμετωπίσουν οι Γεωργοί άλλο πρόβλημα διότι ε, εάν δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τα παράσιτα ε, δεν μπορεί ε, να καλλιεργήσει κανείς ε, κήτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει το παρασιτοκτόνο. Οι μικρές καλλιέργειες συνήθως είναι πράσινοι γεωργοί ε, συνήθως καλλιεργούν ε, κρυθάρι με πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί ε, να τους εμποδίσουμε. Επίσης, εάν έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις τι θα κάνουν αυτές θα ζητήσουν από μια μεγαλύτερη εκμετάλλευση να τους, ε, να συνεργαστούν με μια, μεγάλη εκμετάλλευση η οποία θα τους πει όμως ότι εγώ μπορώ να συνεργαστώ καλύτερα μαζί σας εάν την ε, μία χρονιά καλλιεργείται αποκλειστικά στάρι, την άλλη αποκλειστικά βρώμη. Και... Ε, ο ε, ε, ε, συμβαλόμενος θα πρέπει να συνεχίσει να επισκέφτεται την εκμετάλλευση αυτή. Βλέπω ότι ο Τζοζέ κουνάει το κεφάλι του. Σας υπόσχομαι όμως ότι η μεγάλη εκμετάλλευση θα κάνει καλή συμφωνία με τη μικρή εκμετάλλευση εάν έχει ενιαία καλλιέργεια. Οι μεγάλες καλλιέργειες ούτως ή άλλως συγκεντρώνουν τις καλλιέργειές τους εγώ δεν θέλω να βοηθήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, έχει καλή πολιτική, αλλά εάν ε, θέλετε να λύσετε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να ε, ανεβάσετε τα κατόφλια, να αυξήσετε τα κατόφλια. Αναφέρθηκε η αγρανάπαυση, αναφέρθηκαν οι εστιασμένες περιοχές και το ποσοστό το 70%. Αναφέρθηκε ότι μπορούν να ενσωματωθούν εδώ υπάρχοντα στοιχεία. Υπάρχουν όμως τεράστιες εκτάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο τα λεγόμενα φένζο που καλλιεργούν λαχανικά δεν χρειάζονται την ε, ε, ενιαία ενίσχυση. Τα σούπερ μάρκετ όμως θα τους πούνε ότι μπορείτε να αποκτήσετε την ενίσχυση αυτή θα πρέπει ε, να αφαιρέσουν το 6% των εκτάσεων όμως από την καλλιέργεια. Ε, επίσης τα σίλς είναι καταπληκτικές εκτάσεις. Υπάρχει πολύ μικρή δυνατότητα να, ε, θα πρέπει να αφαιρέσουν πολλά εκτάρια μόνο και μόνο για το μέτρο αυτό. Αυτό πραγματικά δεν φαίνεται να έχει νόημα. Και τελικά ποιο είναι ο στόχο. Στόχο δεν είναι να ελέγξουμε ε, την προμήθεια. Εάν τα κάνουμε όλα αυτά, θα βελτιώσουμε από ό,τι φαίνεται τον καιρό στον κόσμο, το κλίμα. Δεν έχω ακούσει ούτε ένα ε, καλό ε, επιχείρημα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφο Λάιον. Ε, ε, επί δύο-τρία χρόνια θα ε, είναι πολύ δύσκολη η είσοδος των ανθρώπων ε, στη γεωργία και συζητήσαμε τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Υπάρχει ανησυχία ότι μεγάλες επιχειρήσεις θα ζητήσουν ενιαίες ενισχύσεις και ο μόνος τρόπος να εξετάσει κανείς αν είναι επιλέξιμες ή όχι είναι να κοιτάξει κανείς τον τελευταίο του συσυλλογισμό, ο οποίο όμως μπορεί να είναι από πριν δύο-τρία χρόνια. Ε, αυτό λοιπόν ε, σίγουρα θα προκαλέσει σύγχυση. Τέλος, ε, για τη ζάχαρη. Οι προτάσεις αυτές θα ανατρέψουν και τον τομέα των τέφτλων και του ζαχαροκάλαμου. Ο ε, στον τομέα των τεύτλων ε, είναι πολύ νωρί για να έχουμε και άλλη ριζική αλλαγή. Ε, η Βρετανία ήταν ένα από του πιο αποτελεσματικού παραγωγούς, αποδοτικούς παραγωγούς, ωστόσο χάσαμε μεγάλο μέρο τη παραγωγή μα. Δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε ποσοστώσεις για τα επόμενα 6-7 χρόνια και στο Ζαχαροκάλαμο βλέπουν ότι τα τεύτλα βλέπουν απελευθέρωση τη αγορά. και η ενώ οι ίδιοι έχουν ποσοστό σε αυτό θα στοιχήσει 850 θέσει εργασία, μου είπανε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Άγνιου ε, ε, Τζούσεκ κατόπιν ε, Χόφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας συγχαίρω και εγώ και συγχαίρω και όλους για την επανεκλογή τους έχω να πω το εξή. Ακούσαμε ήδη πολλά και γι' αυτό προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Όλοι επιθυμούμε η κοινή αγροτική πολιτική να είναι διαφανής και δίκαιη. Να οδηγήσει δε σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων αγροτών. Όμως, οι αγρότες μας έχουν την εντύπωση ότι δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η νέα πρόταση για τις άμεσες πληρωμές. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα με την ε, νέα πρόταση. Όπως λέει η μελέτη επιπτώσεων της Επιτροπής, το νέο σύστημα και κυρίως για τις νέες χώρες μέλη που έχουν το σύστημα SAP θα σημάνει σημαντική αύξηση δαπανών και γραφειοκρατική επιβάρυνση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να παραταθεί η ισχύ του συστήματος SAP γιατί είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Και σε ό,τι αφορά την όροφη, το capping, στη χώρα μας και στην Τσεχική Δημοκρατία λόγω του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αντίθετοι με το σύστημα αυτό που θα σημάνει αυξημένη γραφειοκρατική επιβάρυνση για αυτές. Και υφίσταται δυσμενή μεταχείριση με τον τρόπο αυτό η εκμεταλλεύση μας. Και σε ό,τι αφορά τώρα το πρασίνισμα της ΚΑΠ, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι εθελοντικά και να προσφέρουν κίνητρα. Αυτό το 7% υποχρεωτικό μέτρο θα σημάνει μεγάλες ζημίες για την ευρωπαϊκή γεωργία. Θα σημάνει άλλωστε περισσότερες επιθεωρήσεις και ελέγχους και άρα πάλι μεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Και σε ό,τι αφορά τον ορισμό του ενεργού αγρότη, Ας δώσουμε κάποια ευελιξία στο εθνικό επίπεδο για να μπορεί να σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας μέλους. Εν συμπεράσματι, θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβασμό για τη νέα πρόταση μεταρρυθμίσεως και δεν είμαι βέβαιος θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ακόμα και εντός των πολιτικών ομάδων. Ίσως περισσότερο μπορέσει να δημορφωθεί συνένεση μεταξύ εκπροσώπων της ίδιας χώρας παρά μεταξύ πολιτικών ομάδων, πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ντόρφμαν και μετά ο Μισελ Νταρντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και από τη μεριά μου για την επανεκλογή σου. Αυτό αποτελεί και σημάδι της ε, καλής δουλειάς των τελευταίων ετών. Πολλά ελέγχθησαν ήδη. Νομίζω ότι μπορώ να συμπληρώσω ορισμένα βέβαια πράγματα. Η μετάβαση από ένα ιστορικό μοντέλο σε μια ε, πρημοδότηση στη βάση της περιφέρειας είναι στην ουσία απαραίτητη. Και ναι μεν ασκείται κριτική σήμερα σε αυτή τη μετάβαση, αλλά θα πρέπει να εξετάσει κανείς ποιος υποστηρίζει τόσο πολύ αυτές τις ιστορικές πρημοδοτήσεις. Είναι αυτοί που απολαμβάνουν σήμερα τέτοιες πρημοδοτήσεις. Αλλά από τη χώρα μου, όπου εξακολουθεί και ισχύει η ιστορική μέθοδος υπολογισμού, έχει, είναι σαφές ότι έχει περάσει ο χρόνος της πλέον. Υπάρχουν απολύτως αδικαιολόγητα και εκτιμένα εκμεταλλεύσεων που όπως είπα δεν έχουν απολύτως καμία δικαιολογία πλέον, καμία ε, δικαίωση, κανένα δίκαιο να λαμβάνουν αυτές τις πρημοδοτήσεις. Και όμως θα κάνουν κάθε τι το δυνατόν ε, για να συνεχίσουν να τις λαμβάνουν, έστω και με πράγματα τα οποία δεν θα εξυπηρετούν την γεωργία. Η ρύθμιση για τους μικρούς παραγωγούς είναι σωστή και είμαι αντίθετος με αυτό που το κύριο Σιλβέστρης προηγουμένως που είπε ότι κάτω από 100.000 δεν θα πρέπει να καταβάλλονται κάτω από 100.000 είναι όμως είναι 37% ε, όλων των εκμεταλλεύσεων στην περιφέρειά μου. Επίσης στην περιφέρειά μου παρόλο που στην Ιταλία είναι περίπου 325 ευρώ, στην περιοχή μου είναι 100 ευρώ και αυτό έχει πάλι σχέση με το ιστορικό μοντέλο ευρώ λοιπόν είναι 100 εκτάρια και 100 εκτάρια για μας στην περιοχή μου είναι μεγάλη εκμετάλλευση. Άρα οφείλει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο το γεγονός ότι μια εκμετάλλευση είναι μικρή δεν σημαίνει ότι δεν ασκεί η γεωργία η οποία είναι στραμμένη προς τις ανάγκες της αγοράς. Και του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα και στην περιοχή μου, την Καρινθία δηλαδή, που είναι αλπικές περιοχές, να τα δούμε αυτά τα πράγματα σε επίσκεψη αντιπροσωπείας και θα μπορέσουμε να τα διαπιστώσουμε επί Για τα μέτρα πρασινίσματος. Εμένα μου προκαλεί την εντύπωση ότι είναι μια απελπισμένη προσπάθεια να βρουν κάτι που να είναι κάπως λογικό. Και ωστόσο τελικά τα αποτελέσματα είναι παράλογα. Και είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με τον κύριο Ανιό που μίλησε προηγουμένως, μάλλον το λέω και εγώ λάθος το όνομά του, το γεγονός ότι υπάρχει η εναλλαγή καλλιεργιών δεν σημαίνει ότι είναι και αγρονομικά ορθή. Εάν δηλαδή κάποιος σπείρει σιτάρι μετά από κρυθάρι και μετά από βίνι, δεν είναι καθόλου ε, λογικό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν οι αγρότες να είναι εκπαιδευμένοι, χρειάζονται αγρονομικές συμβουλές και να τους εξηγήσει κάποιος αν είναι σωστό να καλλιεργούν καλαμπόκι ή στάρι κλπ. Και αυτό το 7% της αγρανάπαυσης ίσως για ορισμένες περιφέρειες να είναι λογικό, για άλλες όχι. Η αυτόματη αγρανάπαυση σε εμά είναι και από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα, διότι δεν γίνεται πλέον αντικείμενο ορθής διαχείρισης ε, το περιβάλλον, το τοπίο εκεί. Επανέρχομαι λοιπόν σε κάτι το οποίο έχω ξαναπεί εδώ και στη διάρκεια συζητήσεων της εκθέσεως DES θα προτιμούσα να συζητήσουμε για την ανάπτυξη των αγροτοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει πολύ περισσότερο σε βελτίωση του περιβάλλοντος, θα είμαστε πλέον αξιόπιστοι στα μάτια των γεωργών και βέβαια πιο ανταγωνιστική. Και τώρα κάτι για τις μειονεκτικές περιοχές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν προκειμένου οφείλει να βελτιωθεί. Οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν γίνει. Περιλαμβάνονται όλα στην πρόταση όπως ήταν στην αρχή και θα πρέπει πάλι νομίζω να εγκύψουμε σε αυτά. qui vous ont été adressés à vous même et aux membres du bureau pour votre Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Ένα θέμα ζήμωσης μεταξύ ημών είναι το θέμα της ανακατανομής των ποσών μεταξύ των κρατών μελών. Δεν ξεκινάμε από, τίποτα, το τίποτα. Στην έκθεση John Lyon εμείς είχαμε βρει μια φόρμουλα συνενετική που έλεγε δίκαιη κατανομή, αυτό δεν σημαίνει ισότιμη αναμονή, α, κατανομή. Στην έκθεση Παρδές ζητούσαμε από την Κομισιόν να μας δώσει στοιχεία, συγκριτικά στοιχεία όπου αναφορικά με το εισόδημα, τις δαπάνες κλπ. για να κάνουμε την κατανομή. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές του βιωτικού επίπεδου μεταξύ των 27, μου φαίνεται δύσκολη σε πέντε χρόνια να έχουμε μία πλήρη αρμονία, αυτός βέβαια είναι ο στόχος που συμμεριζόμαστε και που πρέπει να προσεγγίσουμε. Για το θέμα του greening και της οικοαναιρεσιμότητας. Τι θέλει να πει αυτό. Οι χώρες μας ε, σχετικά με την οικοανερεσιμότητα εφάρμοσαν τις 15 οδηγίες όπως ήθελαν. Άμα δούμε εμείς τον συγκριτικό ε, πίνακα για το πώς εφαρμόζονται, βλέπουμε ότι τελικά στρεβλώσαμε την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των γεωργιών των διαφόρων χωρών μας, διότι δεν είναι παντού ίδιες αυτές οι οδηγίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλη αυτή η ιδέα του greening, που εντάξει να μην είναι τρία μέτρα, δεν είναι πέντε και έξι, και που θα επέτρεπε την εφαρμογή αυτής της εικοναρεσιμότητας όσο το δυνατόν πιο παρόμοια μεταξύ των κρατών μας δεν θα αποτελούσε μια βάση δικαιοσύνης μεταξύ, μια δίκαιη βάση συγγνώμη, μεταξύ των γεωργών μας. Για το θέμα της κατανομής της χρηματοδότησης και η μεταφορά του από τον ένα πυλώνα στον άλλον. Προσοχή! Εάν διάβασα καλά τις προτάσεις του δεύτερου πυλώνα, η Κομισιόν προτείνει και μία διεύρυνση στο δάσος. Έχουμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα, έχουμε τα συνοδευτικά μέτρα των ΚΟΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία, θα επανέλθω αργότερα σε αυτά. Αν κρατήσουμε λοιπόν εμείς τις πιστώσεις για τις μειονεκτικές περιοχές, για όλες τις χώρες θα έχουμε λιγότερα λεφτά για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Πρέπει να έχουμε συνείδηση του πράγματος, πρέπει να το αποφασίσουμε μεταξύ μας. Διότι δεν μπορούμε εμείς να λέμε εντάξει θα κάνουμε παραπάνω εδώ, παραπάνω εκεί γιατί... Ε, και θα κάνουμε παραπάνω παντού. Γιατί αλλιώς θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να ξέρουμε πού στοχεύουμε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου, τα υπόλοιπα τα είπαν άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Μισελ κύριος Γιάρ και μετά ο Νίκολσον. Ευχαριστώ. Ευχές και συγχαρητήρια και από μένα. Έχω σημειώσει τρία-τέσσερα σχόλια. Πρώτο, ας θυμηθούμε τις δικές μας τις αποφάσεις ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό θα πρέπει να εγκρίνουμε την τελική μεταρρύθμιση όταν γνωρίζουμε προς τα που κατευθυνόμαστε με τα δημοσιονομικά. Δηλαδή να κάνουμε τις σχετικές διαβουλεύσεις, να συντάξουμε τα σχετικά έγγραφα, αλλά να μην λησμονούμε γεωρική μεταρρύθμιση, τελική απόφαση και προϋπολογισμός. Όλα αυτά βέβαια είναι αλληλοσυνδεόμενα μεγέθη. Δεύτερη παράκληση, γραφειοκρατία. Έχω την μεγάλη ανησυχία ότι στην προσπάθειά μας να τα κάνουμε όλα δικαιότερα και καλύτερα, ότι θα εισαγάγουμε ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία στο σύστημα. Κάθε λοιπόν φορά που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα, ας φροντίσουμε να μην οδηγήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία με τις προσπάθειες βελτιώσεως. Και γι' αυτό, όπως είπαν και άλλοι πριν, για το πρασίνισμα για παράδειγμα, θα παρακαλέσω τον εισηγητή και αυτός να συνταχθεί με την προσπάθεια να δούμε οι εκμεταλλεύσεις εκείνες οι οποίες ήδη συμμετέχουν σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα να απαλλάσσονται από τα μέτρα του πρασινίσματος. Στην περιοχή μου υπάρχουν πολλοί αγρότες που δεν αντιλαμβάνονται την αξία των προτάσεων του Επιτρόπου για το πρασίνισμα, διότι λένε «Μα όλα αυτά που μας ζητάει τα κάνουμε, τι άλλο θέλει». Επομένως, εκμεταλλεύσεις οι οποίες ήδη κάνουν πράγματα για το περιβάλλον να μην τελικά υποστούν μια δυσμενή μεταχείριση. Πάλι για το πρασίνισμα, τα πράγματα πρέπει να είναι και λογικά και ειδικά για την εναλλαγή καλλιεργιών Το παράδειγμα που φέρνω συχνά όταν ένας αγρότης έχει 50 εκτάρια αρρώσιμη γη, θα πρέπει να χωρίσει την γη του σε τρία μέρη και να καλλιεργήσει τρία διαφορετικά πράγματα. Ο άλλος ο οποίος έχει διάφορα εδάφη μπορεί κάθε χρόνο και στο ίδιο μέρος μάλιστα να καλλιεργεί 70% ε, ε, σιτηρά κάθε χρόνο. Εμείς θέλουμε εναλλαγή καλλιεργιών και βάζουμε τρία, τρία διαφορετικά είδη σε κάθε χωράφι κάθε χρόνο, πάντα τα ίδια. Ευαισθησία δείχνουν οι αγρότες στην περιοχή μου αφενός για την ταχύτερη προσαρμογή. Εγώ προέρχομαι από την Ανατολική Γερμανία, είχαμε πει και παλαιότερα εκτάριο είναι εκτάριο και κάναμε την προσαρμογή σύντομα κυρίως με την επανένωση των δύο Γερμανιών κατανοώ νόμος και τους συναδέλφους από τις νέες χώρες μέλη ότι εδώ χρειάζεται να δοθεί ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα προς την κατεύθυνση μιας προσαρμογής. Εδώ είναι όμως οι αγρότες ιδιαίτερα ευαίσθητοι και σε ό,τι αφορά την οροφή, το κάπινγκ. Εγώ 30 χρόνια, τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής μου Έζησα σε μια χώρα όπου μας επέβαλαν και τι θα καλλιεργήσουμε, πόσα ζώα θα εκτρέφουμε την τελευταία λεπτομέρεια. Γι' αυτό αυτό το κάπινγκ για μας είναι καθαρός κομμουνισμός. Δηλαδή άνωθεν επιβαλόμενες δεσμεύσεις. Ενώ οι αγρότες μας επιθυμούν να μπορούν οι ίδιοι να επιλέγουν με ποιον τρόπο θα διαχειριστούν την εκμετάλλευσή τους. Τελευταίο παράδειγμα που πρέπει πάλι να φροντίσουμε να μην οδηγήσουμε σε μεγάλη γραφειοκρατία είναι ο περίφημος ενεργός αγρότης. Πριν να συγκεκριμενοποιηθούν οι προτάσεις του Επιτρόπου, εγώ έλεγα συχνά ότι η μόνη διάκριση που γνωρίζει τον Γεωργό είναι τεμπέλης Γεωργός, επιμελής Γεωργός. Τώρα έρχομαι και στον ενεργό Γεωργό. Τι είναι αυτός ο ενεργός αγρότης να συνδεθεί λέει με, με το εισόδημα. Εγώ τώρα γράφω την ε, φορολογική μου δήλωση για το 2010 και δεν είμαι και ο τελευταίος, είναι και άλλοι που έχουν ε, αργήσει. Αν λοιπόν είμαι ενεργός αγρότης θα πρέπει να πληρώσω ξανά. Μια φορά ο αγρότης θα είναι ενεργός, μια φορά δεν θα είναι. το εάν ο αγρότης είναι ενεργός ή όχι πρέπει να φαίνεται και από τον τρόπο που διαχειρίζεται τις γέες του, τις εκμεταλλεύσεις του. Και τέλος, να φροντίσουμε να μην βλάψουμε μια πελατεία που δεν έχουμε κανένα λόγο να ε, βλάψουμε. Αντίθετα πρέπει να προστατεύσουμε και τις μειονεκτικές περιοχές. Και εδώ λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε πολύ καλά αυτό τον ενεργό αγρότη, γιατί καμιά φορά λιγότερα είναι εν τέλει περισσότερα. Ευχαριστώ κύριε Γιάχ. Ο Τζιμ Νίκολσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ όσους ε, εξελέγησαν να παρακαλέσω τον κύριο Αγνιού να μην αλλάξει, διότι μόλις συνηθίσαμε πώς είναι. Μόλις τον προσαρμοστήκανε, ε, ε, δεν θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε κάποιον νέο κύριο Άγνιου. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Καπλασάντος, διότι δεν ήμουν εδώ κατά την παρουσίασή του. Ε, άκουσα όμως την συζήτηση και υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δείχνει η συζήτηση αυτή. Πόσο διαφέρουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. άκουσα τα σημαντικά προβλήματα που έχει η κάθε περιφέρεια, η κάθε περιοχή. Και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ε, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή. Όλοι μιλάνε για απλοποίηση. Τίποτα δεν θα απλοποιήσει αυτή η μεταρρύθμιση. Πιο πολλή γραφειοκρατία, πιο πολλά προβλήματα, πιο, πολλές εκμεταλλε... πιο πολλά έντυπα, πιο πολύ, πιο πολύ διοικητικό κόστος. Τα πάντα υπόθηκαν στη συζήτηση αυτή, στις ε, περιφέρειές μας οι γεωργικοί σχολιαστές ε, έχουν γράψει πάρα πολλά. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές για μένα, ότι ε, ένα κουστούμι δεν κάνει για όλους. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στον τομέα αυτόν. Ε, για παράδειγμα, η ενεργή γεωργία είναι διαφορετικός ορισμός σε κάθε περιφέρεια. Πώς θα το εφαρμόσουμε, πώς θα εφαρμόσουμε σχετική διάταξη και το να την εφαρμόσουμε σε μια χώρα και όχι σε άλλη, αυτό θα είναι φιάλτης. Κύριε Πρόεδρε, πριν δύο χρόνια όλοι μιλούσαν για την ε, τροφοδοτική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα για να ταΐσουμε τον κόσμο. Και τι μας λέει η Κομισιόν, ότι θα πρέπει να, ε, ε, ε να έχουμε αγρανάπωση στο 7% των εκτάσεών μας. Μα πόσο τρελός μπορεί να είναι κανείς. Η δουλειά της Επιτροπής μας είναι να βάλουμε λίγη κοινο, ε, κοινή λογική στο μέλλον της γεωργίας. Να μην προσποιούμεθα και να μην συνεχίσουμε κάνοντας τα ίδια που κάναμε πριν 7 ή 10 χρόνια. Τώρα έχουμε τη συναπόφαση. Ε, αυτό είναι εξουσία της Επιτροπής μας ε, και πρόκληση για μας είναι να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά ως ε, μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Διότι κύριε Πρόεδρε, αν δεν το κάνουμε αυτό, οι γεωργοί της Ευρώπης σε κάθε κράτος μέλος θα υποφέρουν. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ας ανταποκριθούμε σε αυτήν. Ευχαριστώ Τζιμ. Σίγουρα, σίγουρα θα πρέπει να δράξουμε όλη αυτή την πρόκληση. Μας δεσμεύει όλους, μας, δίνει μια, αναθέτει μια τεράστια ευθύνη. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά. Οι εισηγητές μας είναι αυτοί που θα πρέπει να προθήσουν τις προτάσεις στην Επιτροπή μας. Τέλειωσαν οι συζητήσεις. Α, δίνω το λόγο στον Διευθυντή Πατσέκο της ε, Κομισιόν και μετά ο καπούλας να μας δώσει τα τελικά σχόλια. Τελευταίο σημείο στο Μισελ Νταντά μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ ε, εγώ και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής σας ε, για τις ενέργειές τους. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας και βρισκόμαστε απολύτως στη διάθεσή σας. Στόχος ε, τώρα δεν είναι να σας παρουσιάσω τις δικές μας ε, θέσεις ε, για τη συζήτηση που μόλις ακούσαμε. Να πω λίγα λόγια όμως. Από την προκατακτική αυτή συζήτηση βλέπω ότι υπάρχει γενική στήριξη για το πλαίσιο. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τις λεπτομέρειες της πρότασης. Και για παράδειγμα όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσει το πρασίνισμα, ποιε θα είναι ε, οι οικολογικά εστιασμένε περιοχές, ποιο είναι ο ορισμό του ενεργού γεωργού. Πολλή δουλειά απομένει ακόμα να γίνει, το αναγνωρίζω αυτό. Προτείναμε να γίνει. Είμαστε διατεθειμένοι εν ευθέτω χρόνο να ε, συζητήσουμε μαζί σας τις ιδέες μας για το πώς θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Δεν είναι όμως εύκολο έργο αυτό. όσον αφορά το πρασίνισμα και τον ενεργό γεωργό να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όσον αφορά το greening, το πρασίνισμα, αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να πούμε ότι οι γεωργοί ωφελούν γενικά την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας σύνδεσμος με τα κοινά αγαθά που προσφέρει η Γεωργία και ακριβώς ε, αυτό μας απασχολεί στο greening. Και όσον αφορά τις οικολογικά εστιασμένες περιοχές, η EFA, προτείνεται αγρανάπαυση 7%. Αυτό το είπαμε από την αρχή και πολύ σαφώς. Οι οικολογικές ε, οι οικολογικά εστιασμένες περιοχές δεν είναι αντικείμενο αγρανάπαυσης. Έχουμε συζητήσει τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, αλλά σίγουρα στοιχεία που σήμερα συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες περιοχές, όπως για παράδειγμα οι φράχτες από θάμνους, ε, όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στις οικολογικά εστιασμένες περιοχές και θα μπορέσουμε έτσι να συμβάλλουμε στο καλύτερο περιβάλλον και στην βιοπικιλότητα. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή μαζί σας. Μία παρατήρηση για τον ενεργό γεωργό. Έχουμε σήμερα έναν τρόπο να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να αποκλείουν μεγάλες επιχειρήσεις από τις άμεσες ενισχύσεις. Μία χώρα μόνο έχει εφαρμόσει το μέτρο αυτό. Μας συζητήθηκε να υποβάλουμε έναν πιο ακριβή ορισμό ώστε να πετύχουμε το στόχο που από τη συζήτηση και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη συμμερίζεστε όλοι. Ε, ότι ο ενεργός γεωργός, όχι η μεγάλη επιχείρηση, θα πρέπει να λαμβάνει τις πληρωμές, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διακινδυνεύουμε το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων. Εάν για παράδειγμα πούμε ότι δίνουμε άμεσες ενισχύσεις σε όλους που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν παράγει και διαθέσει στην αγορά τα προϊόντα τους, τότε ε, παραβιάζουμε ε, κανόνες του ΠΟΕ για ε, το Green Box, για το Πράσινο Ταμείο. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια πολύ λεπτή γραμμή, διότι θέλουμε να πετύχουμε το στόχο που συμμερίζεστε όλοι και ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, φροντίσουμε οι άμεσες πληρωμές μας ε, να ε, θεωρείται ότι επίπτουν στο green box του ΠΟΕ. Δεν είναι εύκολος ο ορισμός. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια και είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για να βελτιώσουμε την πρόταση. Και πάλι κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω και προσλέπουμε στη συνέχεια της καλής συνεργασίας μαζί σας. Ευχαριστούμε την Κομισιόν ε, αδιαμφισβήτητα για αυτό το θέμα του 7% της οικολογικής ε, ε, των οικολογικών εκτάσεων υπάρχουν διάφορες ανησυχίες και το ακούσατε εδώ όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας εκφράστηκε και αλλού σίγουρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην διατύπωση της διότι άμα δημιουργούνται πια τόσο ανησυχίες, τόσες ανησυχίες θα πρέπει κανείς να ξαναδεί την πρόταση. Ο Λουίς τώρα για τελικά σχόλια και μετά ο Μισελ Νταντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για να δώσω το χρόνο στο συνάδελφο Νταντέν να παρουσιάσει την δουλειά του. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν, οι οποίες ε, ε, μου επέτρεψαν να καταγράψω τις τάσεις της Επιτροπής. Εγώ στην αρχή δεν ευχαρίστησα την Κομισιόν για την ε, διαθεσιμότητα, για τη διάθεσή της να συνεργαστεί. Εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα είχα επαφές με τον Επίτροπο και τον Γενικό Διευθυντή οι οποίοι είπαν ότι θα ήταν καλό να έχουμε μία μόνιμη task force ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αυξομοιώσεις ε, και να έχουμε συνεχή παρακολούθηση. Χαίρομαι που υπάρχουν ε, κεντρικά πολιτικά θέματα τα οποία συμπίπτουν με αυτά τα οποία εγώ είχα αναφέρει. Ο συνάδελφος Λάιον έφυγε αλλά έκανε μια πολύ εύστοχη ερώτηση υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα το οποίο δεν φύχτηκε μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι η Κομισιόν διατυπώνει μία πρόταση κατανομής του προϋπολογισμού, ενώ αυτή η πρόταση έπρεπε να είναι αντίθετο, αντίθετη. Δηλαδή πρώτα να οριστούν τα κριτήρια και μετά θα βλέπαμε πώς θα εφαρμοζόντουσαν αυτά τα κριτήρια και πώς θα διαμορφωνόταν η <coughs> ο χρηματοπιστωτικός φάκελος για την κάθε χώρα. Εγώ διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει φοβερό, φοβερή αντίδραση από το κοινοβούλιο δεν υπάρχει φοβερή αντίδραση από το Κοινοβούλιο ούτω ώστε μετά να πάμε μαζικά να τροποποιήσουμε ε, ριζικά την πρόταση. Ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας. Τώρα αν θέλουμε εμείς κάποιον κατάλληλο μηχανισμό προσαρμογής θα πρέπει να το συζητήσουμε και για το παράρτημα 2. Το θέμα λοιπόν θα είναι ένα δύσκολο πολιτικό θέμα, θα ήταν σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας διότι όλα τα κράτη θα θέλανε παραπάνω κονδύλια. Αυτό είναι το βασικό πολιτικό ζητούμενο. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα νομικής νομιμότητας όπως έλεγε ο συνάδελφος Λάιον. Πρόκειται για ένα πολιτικό θέμα πολύ λεπτό. Αυτή ήταν μία πρώτη συζήτηση και εγώ έχω τις ε, γνώμες μου για τα διάφορα σημεία, αλλά θα τίνω προς τη συνένεση. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο ε, ε, να έκανα μια δική μου προσωπική έκθεση αντιτελείωνας 24 ώρες. Εγώ φαντάζομαι ότι όμως ότι το κοινοβούλιο δεν θα την ενέκρινα αμέσως. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας, δεν είναι μία έκθεση η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις δικές μου θέσεις, ούτε και το αντίθετο βέβαια των θέσεων μου. Πρέπει να βρούμε μία συνένεση για να έχουμε ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια για να εμφανιστούμε ισχυροί γύρω από τους ουσιαστικά ζητήματα εγώ θα εργαστώ προς αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε να συσπυρώσω όλες εκείνες τις τοποθετήσεις που θα με οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση της κοινή θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ, Λουίς. Τελευταίο σημείο για την μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγορών. Ο Μισελ Νταντά έχει το λόγο. Μισελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να τα πω γρήγορα θα πω ότι μεθοδολογικά ακολούθησα την ίδια μέθοδο με τον Λουίς. Οπότε και εγώ βρίσκομαι σε μία φάση διαβουλεύσεων, μαζεύω γνώμες και πραγματογνωμοσύνες. Ένα αίσθημα καταρχήν. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το κείμενο για την ΚΟΑ έχει περάσει σε δεύτερο, σε δεύτερο πλάνο γιατί συζητάμε κυρίως το θέμα του greening και το θέμα της κατανομής των ενισχύσεων. Πολλές φορές η Επιτροπή μας εκφράστηκε σχετικά με την ανάγκη να εφαρμόσουμε διάφορα μέσα διαχείρισης και ρύθμισης των αγορών. Και αυτό το κείμενο είναι και ο φορέας όλης αυτής της ουσίας. Σχετικά με το κείμενο το ίδιο να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο ή τρία σημεία. Για τα μέτρα διαχείρισης των αγορών. Έχουμε μια σειρά διατάξεων και μέτρων, μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τον ίδιο τον Γεωργό μέσω της ασφάλειας, της οργανώσεις των, αγρι... των ε, γεωργών, οι οποίες ε, διαμορφώνουν ε, στους κόλπους τους ε, ασφαλιστικά ταμεία, ενίσχυση για την ιδιωτική αποθήκευση που είναι κάτι το πιο συλλογικό και μετά φυσικά έχουμε και το δίκτυο ασφάλειας που είναι η κρατική ενίσχυση. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπόθηκαν όλα σαφώς, κυρίως για την ενίσχυση στην ιδιωτική αποθήκευση. Η πρόταση στο άρθρο 17 προτείνει να ανοίξουμε την, την ιδιωτική αποθήκευση σε ένα νέο κριτήριο, το οποίο διεκδικήσαμε σε προηγούμενες εκθέσεις. Και πρόκειται και για μια διεκδίκηση των επαγγελματίων. Έχει να κάνει και με την εξέλιξη των τιμών. Λέει να κολλήσουμε όμως και στην εξέλιξη του τομέα. Όταν συγκρατιούμε τις τιμές αλλά οι επιβαρύνσεις τα έξοδα ε, ε, αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενεργοποιήσουμε την ενίσχυση για, στην ιδιωτική αποθήκευση. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν βρίσκεται εκεί η ουσία της έκθεσης. Η ουσία είναι η προσφορά που δίνεται στον παραγωγό να ενισχύσει την οργάνωσή του και αυτό μας επιτρέπει να γράψουμε αυτό το οποίο λέει το άρθρο 42 της Συνθήκης της Λισαβόνας όπου λέει ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να παρεκκλίνουν στο άρθρο 101 για τους κανόνες του ανταγωνισμού. Όταν εγώ ακούω τους κύκλους της Κομισιόν και του Επιτρόπου, όλα είναι εφικτά. Εγώ προσπαθώ λοιπόν να μαζέψω όσο το δυνατόν περισσότερα παραδείγματα από τις διάφορες χώρες όπου οι οργανισμοί ανταγωνισμού παρενέβησαν για να σταματήσουν ενώσεις γεωργών. Δηλαδή από τα λόγια στις πράξεις ε, έχουμε δύο κόσμους ε, απόσταση. Το πιο φοβερό παράδειγμα είναι αυτή η 37 παραγωγή μια ποικιλία μήλων όπου η 31 είναι οργανωμένοι σε μια ομάδα παραγωγών οπότε η αρχή κατά το, ε, η προστασία του ανταγωνισμού τους κάνει μήνυση για δεσπόζουσα θέση. Αλλά δεσπόζουσα θέση σε ποιο κλάδο, στα μήλα, στα φρούτα, πού. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να παρέμβουμε και θέλω να υποβάλω προτάσεις όχι για να εξελιχθεί το δικαίωμα στον ανταγωνισμό αλλά για να διευκρινιστεί να διευκρινιστούν ορισμένοι όροι και ορισμένα εφαρμοστικά πεδία. Το θέμα της δεσπόζουσας θέσης, ε, της αγοράς αναφοράς, του ορισμού των συμφερόντων του καταναλωτή. Αυτά πρέπει να τα διευκρινίσουμε στο κείμενο για να αποφύγουμε αύριο να έχουμε μερικοί, και χρησιμοποιώ τον όρο, μερικές α, ε, αλαφρόμυαλες ερμηνείες των κειμένων. Πρέπει να δούμε επίσης τις αναφορές ε, στις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης ε, και στα άλλα ζητήματα που αφορούν στο θέμα της ε, ε, εκπροσώπησης των παραγωγών. Έχουν, από αυτά όμως εξαρτάται και το άλλο κείμενο το οποίο διαπραγματεύεται ο πρόεδρος για τις αβεβαιότητες σχετικά με τη συμπερίληψη ή μη του κείμενου κειμένου του πακέτου ευθυγράμμισης, συγγνώμη, στο κείμενο. Έτσι εργάζομαι, αναλύω όλα τα στοιχεία και βλέπω ότι, γίνανε, ότι έπεσε ψαλίδι στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Ε, μπορεί κανείς να μαντέψει προς ποια κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι η δουλειά μας θα μπορούσε να αποκαταστήσει μέρος των όσων ε, περικόπηκαν διότι όπως ε, είπαμε και άλλες φορές το δικαίωμα του ανταγωνισμού είναι εκεί για να προστατεύει χείρες και ορφανά, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τον παραγωγό. Γκαρσία Πέρες και μετά Ραντς Γκαρσία ή Ράτσε πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επαναλάβω και εγώ τα συγχαρητήρια τόσο στον Πρόεδρο όσο και στους υπόλοιπους ε, του Προεδρείου. Σύμφωνο με τον εισηγητή σχετικά με την ΚΟΑ ότι σίγουρα στην ε, ολική συζήτηση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ το θεμελιώδες είναι όσο, ε, όσο έχουν να κάνουν με την καταμονομή των διαφόρων ταμείων αλλά πρέπει να δούμε όμως και την πραγματικότητα το τι μας ζητάνε οι παραγωγοί μας οι οποίοι λένε ότι η άμεση βοήθεια δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους ότι χρειάζονται άλλα μέτρα για την στήριξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε από κοινού και εις βάθος. Ρωτώ, ρωτώ και εκφράζω και μία αμφιβολία. Λοιπόν, ρυθμίσεις των αγορών, ποσόστοση για της ζάχαρης και δικαίωμα φύτευσης. Πολλές φορές έθεσα το ερώτημα και το ξανακάνω. Εγώ πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες να διατηρηθεί η ποσόστοση ε, καλλιέργεια ζαχαρότευνων στο 2020 με όπως εκφράστηκε και η έκθεση DES και στην ίδια γραμμή θα πρέπει να θέσουμε και τη θέση της Κομισιόν σχετικά. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα φύτευσης για τα ζαχαρότευκλα αλλά και για τους αμπελώνες είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια θα είναι η γραμμή στην οποία στοχεύει το Κοινοβούλιο. Τώρα, αμφιβολία, ερώτηση. Για την διόρθωση της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 106 ως 108 που διορθώνουν την προσφορά με τις ανάγκες της αγοράς, τι γίνεται με τους γαλακτοπαραγωγούς. Ή τις διατάξεις που έχουμε εδώ ή τις διατάξεις που ισχύουν στο γαλακτοκομικό πακέτο. Γιατί συζητάμε τώρα και το θέμα της ποιότητας και του ελέγχου των, των ποσοτήτων. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξαναδούμε αυτό το ζήτημα και να το ξεκαθαρίσουμε. Ποια θα είναι η διαφορά των δύο διατάξεων. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής μπορεί να μου απαντήσει ή κάποιος από την Κομισιόν σχετικά. Ευχαριστώ Ιράτσε. Έραντς Γκαρσία και μετά ο Αντιπρόεδρος Μποβέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια που πριν δεν σας τα έδωσα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε εδώ τρία στοιχεία για την, κοινή, για, για την ΚΟΑ. Ο ρόλος των οργανώσεων των παραγωγών σε αυτή την ΚΟΑ. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ένα πράγμα και μετά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Εξηγούμε. Φαίνεται ότι βασίζονται στις οργανώσεις των παραγωγών για την ε, διαχείριση των ΚΟΑ θέλουν να δημιουργήσουν διακλαδικές οργανώσεις όλους τους τομείς για να ενισχύσουν τους κρίκους της τροφιμικής αλυσίδας και υπάρχει μετά το θέμα όμως της νομικής ανασφάλειας και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Θα έπρεπε να οργανωθούμε ούτω ώστε οι αρχές του ανταγωνισμού ε, στα κράτη-μέλη να μην πνίγουν τις πρωτοβουλίες των ε, γεωργών. Εμείς είδαμε τέτοιου είδους, ε, είχαμε τέτοιου είδους ανασφάλειες ε, στην ε, ελαιοπαραγωγή, στο ελαιόλαδο, συγγνώμη. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν εξαιρέσεις ούτως ώστε η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή να μην χτυπάει, να μην πλήττει τον πρωτογενή τομέα. Τώρα, η Κομισιόν τι κάνει. Εδώ μας προτείνει απαγοητευτικά πράγματα, ενώ καταργεί όλα όσα υπήρχαν προηγουμένως με αυτά που μας προτείνει. Αυτά τα οποία είχαμε εμείς ε, για σημαντικές υποθέσεις όπως, ε, ε, ε, όπως ε, τους τροφιμικούς συναγερμούς που ζήσαμε όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι το Εκόλι. E. Προτείνει δύσκολα πράγματα που δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Θα έπρεπε να έχουμε ένα μηχανισμό κρίσης στο εσωτερικό της ΚΑΠ. Και όχι να περιμένουμε πλειοψηφίες στο Συμβούλιο που μπορεί να μην τις πετύχουμε ή οτιδήποτε άλλο. Θα έπρεπε να έχουμε επίση έναν μηχανισμό γρήγορης επέμβασης όταν έχουμε κάτι το οποίο πλήττει διάφορα κράτη-μέλη. Μπορεί να υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να, πάμε, να φτάσουμε αργά και αποτελεσματικά, αλλά υπάρχουν προβλήματα σε στα νοπά, όπως τα οπορολαχανικά, όπου χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Χρειάζεται επίσης αφήσα λύση για τις κρίσεις στο ελαιόλαδο. Συγγνώμη που το ξαναλέω τρίτη φορά με το ελαιόλαδο, αλλά εδώ και χρόνια αυτός ο τομέας ζητά μία ενημέρωση των τιμών αναφοράς που να απολευθερώσουν την ιδιωτική αποθήκευση. Λοιπόν, οι τιμές είναι εξωπραγματικές σήμερα. Θα έπρεπε να τους προσαρμόσουμε με την τωρινή κατάσταση της αγοράς και η πρόταση της Κομισιόν δεν απαντάει σε αυτό το αίτημα του κλάδου που είναι σωστό. Τελευταίος ομιλητή είναι ο κύριο Μποβέ. Εάν θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο, παρακαλώ κάντε μου ε, ε σημάδι. Μερικές παρατηρήσεις. Ο Μισελ Νταντάν πολύ καλά ανέφερε ποια είναι η βούληση. Η τελική τοποθέτηση όμως για το, για το ψαλίδισμα τη θεωρώ ακόμη πιο σωστή διότι είναι πραγματικά συναφής και δεν φύγει την ουσία, δεν προχωράει μέχρι βάθους. Εγώ πιστεύω με το κείμενο όπως μας προτείνεται σήμερα, η Κομισιόν προσπαθεί όπως μπορεί να λύσει το πρόβλημα της διακύμανσης των τιμών, χωρίς όμως να δίνει λογικές λύσεις για να καταφέρει να λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, προσπαθούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση παίζοντας τους πυροσβέστες, χωρίς όμως να αποφεύγουμε την... Ε, να ανάψει πυρκαγιά. Αφήνουμε τα πάντα στην απορρίθμιση. Το γάλα, τα ζαχαραότεφλα, το θέμα των δικαιωμάτων φύτευσης, όλα αυτά τα, τα απογυμνώνουμε τομέα τον τομέα ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η οργάνωση όλων αυτών των κλάδων οδηγεί στην αποφυγή διακύμανσης των τιμών. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίζουμε μόνο συνολικά το πρόβλημα και μερικώς και κλαδικά πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Τώρα υπάρχει το θέμα διαχείρισης της κρίσης, της ρήτρας διαταραχής, υπάρχει και το θέμα υποστήριξης στα ασφάλιστρα. Εγώ εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν και αναρωτιέμαι μήπως διαφεύγουμε από το ρόλο μας είναι ρόλος της Ευρώπης μέσα από τον προϋπολογισμό της ή των πολιτών μέσα από τους φόρους τους να χρηματοδοτούν τις, ασφ... ασφάλειες. Δηλαδή, εμείς μέσα από τη χρηματοδότησή τους ε, ιδιωτικοποιούμε ε, τις ασφάλειες. Αυτοί τι συμφέρον έχουν, έχουν να χειροτερεύει η κρίση για να βγάλουν λεφτά. Ίσως να κάνω εδώ μια καρικατούρα, αλλά βλέπουμε εδώ το παραδειγματικό κακό μέτρο το οποίο δεν έχει καμία ειφορία. Πέρα από ένα όριο ε, ε, ε, μεγέθους παραγωγής. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη και από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τις ιδιωτικές ασφάλειες. Μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα στοιχεία. Για μένα το σημαντικό ήταν να τα πω αυτά ε, για την ανάγκη να διατηρήσουμε διαχειριστικά μέσα και να επιτρέψουμε ουσιαστικά στους γεωργούς να συμμετέχουν στην διαχείριση της ε, όλης αλυσίδας ε, παραγωγής και όχι ευκαιριακά όπως γίνεται σήμερα. Ε, είχε υποθεί ότι η Κομισιόν ήθελε να εργαστεί περαιτέρω για, να, για το θέμα των τιμών, για να διαπιστώσει τα περιθώρια κέρδους των μεγάλων αλυσίδων διανομής, των μεσαζόντων κλπ. Αλλά δέστε τι γίνεται αν εμείς ε, θέλουμε να προχωρήσουμε μέχρι τέρμα τη συζήτηση, θα πρέπει να τακτοποιήσουμε όλο το τομέα της διαχείρισης για να έχουν σωστές δίκαιες αμοιβέ οι γεωργοί και όχι να μειώνουμε μόνο το θέμα της υπεραξίας στην τροφιμική αλυσίδα. Ο κύριος Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Νταντάν για την παρέμβασή του. Θα προβώ σε ανταλλαγή απόψεων μαζί του ως εισηγητή του, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σίγουρα θα υπάρξουν βελτιώσεις γιατί Στη γεωργία υπάρχει αβεβαιότητα και αναστάτωση στις τιμές. Χρειάζεται μια σειρά από μηχανισμούς που θα προταθούν άλλωστε. Βέβαια, για ορισμένα από τα μέτρα δεν είμαι βέβαιος πώς θα υλοποιηθούν. Τώρα έχω να κάνω δύο σχόλια. Η Κομισιόν μας επιβάλλει τον προϋπολογισμό και ορισμένες χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα που έχουν σχέση και με άλλους στόχους, όχι μόνο με την κοινή αγροτική πολιτική. 3,9 δισεκατομμύρια για τα εγγύησεως. Επίσης για την επισητιστική βοήθεια. Αυτά πρέπει να εγγράφονται στον προπολογισμό του πρώτου πυλώνα, όπως γινόταν και στο παρελθόν. Και κυρίως όταν πρόκειται για την επισητιστική βοήθεια, όπου γνωρίζουμε ότι δύο μεγάλες χώρες μέλη της Ενώσεως έχουν εκφράσει δισταγμούς για την εφαρμογή του μέτρου μετά το 2013. Τι θα γίνει με το ποσό αυτό εφόσον διατηρηθεί η αντίσταση. Πρέπει να δούμε και πώς θα χρησιμοποιηθεί το νέο αποθεματικό εάν δεν περιλαμβάνεται στον πρώτο πυλώνα. Αυτά επιθυμώ να τα κατανοήσω περισσότερο και γι' αυτό θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες και από τον εισηγητή αλλά και από, το, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γεια. Ευχαριστώ. Ένα πρόβλημα όπου δεν γνωρίζω τη λύση, αλλά χρειαζόμαστε μια λύση και εφόσον πρόκειται για τιμές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τους μηχανισμούς της αγοράς. Το παρελθόν κατέδειξε ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε την αντίφαση αυτή, όπου αφενός έχουμε πολλούς μετέχοντες στην αγορά, έχουμε μια μεταπληκτική βιομηχανία σε βάση μικρής εκμεταλλεύσεως και πολύ συγκεντρωμένο εμπόριο στη Γερμανία τουλάχιστον. Και αυτό οδηγεί εν τέλει στο εάν έχουν αρχίσει να πέφτουν οι τιμές και γίνονται όλο και χειρότερες για τους ε, αγρότες θα έπρεπε ο μηχανισμός της αγοράς να οδηγήσει σε μικρότερη παραγωγή, μικρότερη προσφορά επομένω και άρα αύξηση των τιμών. Δυστυχώς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπει ο αγρότης την τιμή να πέφτει και παράγει περισσότερο γάλα για να αναπληρώσει το εισόδημά του. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τώρα να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της αγοράς. Και πρέπει βέβαια να τροποποιηθούν σχετικά τα νομοθετικά κείμενα. Αφενό χρειαζόμαστε βέβαια κινήσεις αγροτών πρέπει να είναι μεγάλες και ισχυρές. Οι δεμοί δεν πρόκειται να βοηθήσουν. Τι να κάνουμε να, με 30 οργανώσεις γαλακτοπαραγωγών στην Ευρώπη οι οποίες θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεύτερο, πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε και προβλέψεις για την αγορά και να δίνουμε και συστάσεις για την παραγωγή. Και αυτά δεν θα πρέπει να θεωρηθούν όμως ότι είναι συμφωνίες για τις τιμές, καρτέλ δηλαδή, που στη Γερμανία απαγορεύονται, διότι στην Γερμανία εμείς εννοούμε πάντα συμφωνίες για τις τιμές όταν αυτές κινούνται προς τα πάνω, ενώ θα χρειαστούμε και άλλες περιπτώσεις να προβλέπονται. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Και αν είχαμε τις ισχυρές αυτές οργανώσεις των αγροτών, θα έπρεπε αυτές να μπορούν να κάνουν και δεσμευτικές συστάσεις. Θεωρία βέβαια αυτό για τις τιμές. Και τρίτο, εδώ καλούμαστε εμείς να παίξουμε ένα ρόλο, η πολιτική δηλαδή, πρέπει να βοηθήσουμε και χρειαζόμαστε βέβαια εκεί και την βοήθεια της παρέμβασης, της αποθήκευσης δηλαδή. Όταν η αγορά αναστατώνεται πρέπει να μπορούμε να παρεμβαίνουμε πολιτικά και να μπορούμε να αφαιρούμε από την αγορά προσωρινά ένα μέρος της προσφοράς ώστε να επαναλειτουργήσει ο μηχανισμός αγοράς. Αυτό βέβαια είναι απλό ιδέα, δύσκολο στην υλοποίηση. Πάντως πρέπει να δώσουμε με κάποιο τρόπο θάρρος στους γεωργούς, να αλλάξουμε δηλαδή τις ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν οι παραγωγοί, να μπορούν να προκαλούν αλλαγές στην αγορά χωρίς αυτό να θεωρείται ότι πρόκειται για απαγορευμένο καρτέλ, δηλαδή για ε, συμφωνημένες αυξήσεις των, αγορο... των τιμών. Οι αγρότες μας λοιπόν πρέπει να μπορούν να ζήσουν από το εισόδημα της παραγωγής τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καλές και σταθερές τιμές. Και αν είχαμε τέτοιες καλές και σταθερές τιμές, δεν θα χρειαζόταν καν να συζητούμε και να διαφωνούμε για τις άμεσες ε, ενισχύσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον και μετά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Θα είμαι σύντομο. Εμείς ελέγχουμε τον παραγωγό στην Γεωργία. Ελέγχουμε τον μεταποιητή, αλλά ο ελέφαντας είναι εκτός εθούσης και αυτός είναι ο λιανοπολιτής, που αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί το λιανικό εμπόριο είναι τόσο ισχυρό που μπορεί αυτό εν τέλει να αποφασίσει και θα είναι που θα λάβει ο παραγωγός και ο μεταποιητής δεν το έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα η Επιτροπή, η Κομισιόν. Διαχείριση των τιμών. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί το 2007 και 2008. Η Κομισιόν αντέδρασε με καθυστέρηση και όταν αντέδρασε εν τέλει έκανε λίγα πράγματα και με μεγάλη καθυστέρηση. Και πολλοί γαλακτοπαραγωγοί επλήγησαν σοβαρότατα λόγω αυτή τη καθυστέρησης. Όταν η Κομισιόν τα έκανε αυτά, λύθηκαν τα προβλήματα βέβαια στον γαλακτοκομικό τομέα. Αλλά αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή χρειαζόμαστε καλή ανταπόκριση. Η ανταπόκριση αυτή δεν μπορεί να είναι αργή, διότι το πρόβλημα υπάρχει και πρέπει κανεί να κινηθεί για την επίλυσή του το δυνατόν συντομότερο. Άρα πρέπει να έχει κανεί την εργαδιοθήκη του τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γι' αυτό και αυτό είναι που πρέπει να, έχουμε στη διάθεσή μας. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την παρέμβαση, τότε βέβαια προκύπτει σημαντική κρίση και έχουμε στα χέρια μας ένα βαρύτατο πρόβλημα. Τα περί της ε, συσκευασίας των χαρακτοκομικών μάλλον συγγνώμη, τη δέσμη των, των μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα συζητηθεί στο Στρασβούργο και θα απαντήσει η Κομισιόν και στην ερώτησή σας. Εγώ συμφωνώ με τις ανησυχίες του Ζωζεμποβέ για την υπόθεση της ασφάλισης. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει δηλαδή η κατεύθυνση που έχουμε πάρει για τα θέματα ασφαλίσεως. Ήμουνα πρόσφατα στις Ηνωμένε Πολιτείες και ρωτήσαμε κατά επανάληψη τι κάνετε εσείς οι Αμερικανοί δηλαδή και μου είπαν ε, ασφαλίζετε το σπίτι σας, ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας, έτσι δεν είναι. Γιατί να μην ασφαλίσετε και την σοδιά σας. Απλά πράγματα είναι αυτά. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε δημόσια χρήματα για αυτό το λόγο. Πρέπει να δούμε πού πάει, από πού έρχεται η υπόθεση αυτή και ποιο βάρος θα επιβάλλει στους γεωργούς. Στην Αμερική λοιπόν υπάρχει λύση αυτή. Βλέπω και μας έρχεται και μας. Αλλά χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε και στην Επιτροπή Γεωργίας, διότι δεν πρόκειται να φύγει από μόνο του και ίσως χρειαστεί λοιπόν να εγγύψουμε σε αυτό. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Νταντέν για την εισήγησή του που έθιξε ένα σημαντικό θέμα, δηλαδή της ενισχύσεως των οργανώσεων παραγωγών και άλλοι βουλευτές βέβαια έθιξαν το θέμα. Συμφωνώ ότι αφενός οφείλει να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών, να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους θέση καθώς βεβαίως ταυτόχρονα να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες του ανταγωνισμού. Πρέπει να είναι και εύλογοι και ισορροπημένοι. Και συμφωνώ με τον κύριο Νίκολσον που είπε τώρα στο τέλος ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι είναι υπερβολικά μεγάλη η δύναμη του μεγάλου εμπορίου και βαρύνει πολύ και στο εισόδημα των παραγωγών και πρέπει να επιτύχουμε ώστε να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία για το θέμα των κρίσεων, σύντομα. Θα θέλαμε να υπάρξει μια διπλή απάντηση. Αφενός βέβαια ταχεία ανταπόκριση. Αυτό είναι όντως σημαντικό. Εμείς την τελευταία ωστόσο κρίση αντιδράσαμε γρήγορα. Και έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα εργαλεία και ενίσχυση των εργαλείων μας για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα αποθεματικό κρίσιος. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι το εξή. Ευτυχώ δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να αντιμετωπίζουμε σοβαρές κρίσεις. Όταν δεν έχουμε σημαντικές κρίσεις λοιπόν οδηγούμαστε σε ένα δημοσιονομικό ε, πλεόνασμα όπου μπορούμε να το εντάξουμε τον βασικό μας προϋπολογισμό, ας πούμε έτσι. Με ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όταν το χρειαζόμαστε, βέβαια με επίγουσα διαδικασία όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο. Εν τέλει δύο λόγια για την ρύθμιση της αγοράς. Τέθηκε το θέμα ήδη από ορισμένου ευρωβουλευτές για τις ποσοστώσεις της ζάχαρης καθώς και για τις ποσοστώσεις του γάλακτος και για τα, για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελιών. Για τη ζάχαρη νομίζουμε ότι ο τομέας έχει πια αρκετά ενισχυθεί και είναι ανταγωνιστικός, επαρκώς ανταγωνιστικός διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, ότι φέτος το γεγονός ότι διατηρούμε τις ποσοστώσεις μας θέτει σε μια θέση όπου έχουμε μια καλή παραγωγή ζάχαρης, υψηλή, έχουμε ωστόσο τη δυνατότητα να εξαγάγουμε την υπερβάλλουσα παραγωγή ζάχαρης. Και αυτό λόγω του ότι διαθέτουμε ποσοστώσεις. Μπορούμε δηλαδή να επισημάνουμε ότι ορισμένες φορές οι ποσοστώσεις μπορούν να δώσουν μια ψευδέστηση ότι προσφέρουν μια έξτρα ασφάλεια στον τομέα, αλλά δεν εμποδίζουν τον τομέα να συμμετέχει στις παγκόσμιες αγορές, στην αύξηση δηλαδή, να ανταποκρίνεται στην αύξηση της ζήτησης δηλαδή, παγκόσμια. Και αυτό μπορεί να το πράξει ο τομέας της ζάχαρης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Προεδρεύων, ο εισηγητής κ. Νταντάν. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας που στράφηκαν γύρω από το θέμα του δικαίου του ανταγωνισμού. Δεν πρόκειται μόνο όπως λέει το κείμενο να επιτραπεί στους ε, παραγωγούς να οργανωθούν αλλά και γιατί ε, για να κάνουν τι. Διότι το ψαλίδι στο κείμενο έχει οδηγήσει στο ότι να είναι πολύ περιορισμένο το τμήμα που είναι για τις οργανώσεις των παραγωγών. Πρέπει επομένω οι τομείς να μπορέσουν να οργανωθούν. Αλλά πρέπει να πει κανείς ακριβώς μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Ορισμένοι από εσά είπατε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνο εργαλεία για να ρυθμίζουμε τα μετά, τα εκ των υστέρων, αλλά πρέπει να υπάρχει και απριόρι ρύθμιση με τις επαγγελματικές οργανώσεις και βέβαια με τη δυνατότητα της ίδρυσής των. Για τις ποσοστώσεις πρώτα για τη ζάχαρη, σημειώνω ότι στον τομέα δεν συμφωνούν όλοι οι συνομιλητές μου. Στις διαβουλεύσεις που κάνω επί του παρόντος, αυτές μου δείχνουν ότι ο τομέας στρέφεται περισσότερο σε μια κατάσταση χωρίς ποσοστώσεις, αλλά έχει ανάγκη ακόμα από 3-4 χρόνια μέχρι ότου φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό ζητεί, δηλαδή να φτάσει μέχρι το 2019-20 με τις ποσοστώσεις των ε, τεύτρων κλπ. Για το δικαίωμα φυτεύσεως, πολλοί έχουμε τοποθετηθεί δημοσία για το θέμα αυτό. Εγώ είπα ότι θα επαναφέρω την προοπτική του δικαιώματος φυτεύσεως ε, αμπελιών δηλαδή στο κείμενό μου είναι ζήτημα τώρα για το ζήτημα της ασφάλισης συμφωνώ με ορισμένες παρατηρήσεις που έγιναν και οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν τους ε, παραγωγούς τους για να περάσουν τις δυσκολίες αυτές αν δείτε πώς ασκείται η αμερικανική πολιτική είναι πραγματικά ένας από τους μεγάλους τομέας ενίσχυσης των αγροτών. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Η συζήτηση που θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες θα βοηθήσει να ξεκαθαριστούν οι θέσεις. Εγώ πάντως θα χρειαστώ τις γνωμοδοτήσεις σας, τις γνώμες σας και βέβαια και απέναντι στην Επιτροπή υπάρχουν ορισμένες κριτικές αλλά οι προτάσεις είναι ακόμα πολύ άριθμες για την ρύθμιση εξακολουθώ να μην βλέπω εξελιγμένες προτάσεις που να προτείνουν εναλλακτικούς μηχανισμούς. Ευχαριστώ, λέει ο Προεδρεύων. Κυρίε και κύριοι, μπήκαμε σε ένα νέο στάδιο πλέον σε βάθος συζητήσεως της, ε, του κειμένου. και για τις άμεσες ενισχύσεις, άμεσες πληρωμές και την κοινή οργάνωση της ε, αγοράς. Νομίζω ότι αξίζει να σκεφτούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά σε αυτό, οι πληρωμές ή ο κοινός μηχανισμός αγοράς, η κοινή οργάνωση αγοράς. Και η διάρθρωση της παραγωγής, δηλαδή το τι παράγουμε, και δεύτερο η δομή των εκμεταλλεύσεων είναι σημαντικά και αυτά χρειάζονται βέβαια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μηχανισμών στήριξης. Υπάρχει και μια ερώτηση ακόμα που θα τεθεί να ρωτήσουμε δηλαδή τους ίδιους τους αγρότες για την άποψή τους για τις δημογραφικές αλλαγές και το πώς θα εξελιχθούν στην Ήπεθρο. Σήμερα γιορτάζουμε την πεντηκοστή επέτειο της ΚΑΠ, μιας πολιτικής η οποία έχει πλέον όγκο εμπειριών και αυτές οι εμπειρίες πρέπει να αναλυθούν. Οι καιροί αλλάζουν μεν και οι εξωτερικοί παράγοντες γίνονται όλο και σημαντικότεροι, παρόλα αυτά μπορούμε να συναγάγουμε πλήθος συμπέρασμάτων βασισμένοι στην πύρα αυτή. Εν τέλει θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγητές, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και όλες και όλους που συμμετέσχατε σήμερα στη συζήτηση. Αύριο θα συναντηθούμε στην ίδια αίθουσα από τις 9 μέχρι τις 10 συντονιστές. Στις 10 θα αρχίσουμε την συνεδρία της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ.